Αγαπητοί συναδελφοί, καθίστε παρακαλώ. Καλό θα ήταν να καθίσετε παρακαλώ τώρα, γιατί έχουμε πολλές ψηφοφορίες και μετά έχουμε και άλλη δουλειά. Right, I've just been just checking how long we have. We've officially got half an hour for the votes, which I don't think is long enough. Λοιπόν, μισή ώρα προβλέπετε για την ψηφοφορία, ελπίζω να μας στάσει. Πρώτη έκθεση, νέα συμμαχία για την επισητιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Η Μαρία Σιγήτρη έχει το λόγο. Μαρία Χαμπουχ. Ευχαριστώ πολύ, Λίντα. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι όλους τους κοιόδης για την καλή συνεργασία. Νομίζω ότι την έκθεση την κάναμε πολύ καλή. Δεν θα θέλω να καθυστερήσω την ψηφοφορία. Να πω μόνο ότι στην παράγραφο 14, τροπολογία 74, αυτή θα ψηφιστεί αν, αυτή θα καταπέσει αν περάσει η συμβιβαστική που το ελπίζω. Αλλά υπάρχει κάποιο θέμα με τις μεταφράσεις σε ορισμένες γλώσσες Θέλω να πω στους συναδέλφους ότι στα αγγλικά, στην αγγλική μετάφραση, ε, είναι λίγο πιο ελεύθερη μετάφραση. Ευχαριστώ. It was tabled in French. Στα γαλλικά μου λένε ότι έχει υποβληθεί. Δεν έχω τα γαλλικά μπροστά μου, οπότε δεν μπορώ να πω κατά πόσο τα αγγλικά και τα γαλλικά. Θα το κοιτάξουμε πάντως αργότερα για να δούμε την τεχνική αυτή πτυχή. Πάντως τα γαλλικά είναι το πρωτότυπο. Αυτό θα καθορίσει. Ωραία. Λοιπόν, για να κάνουμε μια δοκιμή για την ψηφοφορία, δηλαδή βάλτε τις κάρτες σας, πατήστε ένα κουμπί, να δούμε κατά πόσο δουλεύει το μηχάνημα. Ψηφίσατε όλοι. Ένας λείπει. Ο κύριος Πόγκα. Α, Εκεί είσαστε, εντάξει. Ωραία, λειτουργεί. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Ευχαριστώ Μαρία για τις διευκρινήσεις σου. Αρχίζουμε λοιπόν με τη νέα συμμαχία για την επισητιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Τροπολογία 33. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά. Να ελέγξουμε για τη 41, άμα θέλετε. Θα ελέγξουμε, εντάξει, για τη 41. Ελέγχουμε η ηλεκτρονικά, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε την ίδια πλειοψηφία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε για την 59 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της φοφορίας. Εγκρίθηκε. 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Εξήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 72. Υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 72. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε σαφώς. 73 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 74. Όχι. Καταπίπτει. 75 Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 77. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 88 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 89. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά,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 κατά, αποχές. Το ΕΛΚ δεν αντιδράει, οπότε δεν ξέρω. Ωραία, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. 96 και 97 μαζί. 96 και 97 μαζί. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρα στις φοφορίες. Κατά. Απορρίφθηκε. 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 100 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 101 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 102 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 103 υπέρ. Κατά αποχές θα ελέγξουμε για την 103. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 104 Εγκρίθηκε αυτή. 105 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 108 πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε καλύτερα. 111, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες, απορρίφθηκε. Με διαφορά. 112. Υπέρ, κατά, αποχές,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 μία-μία τότε και θα δούμε αν κάποιες μπορούμε μαζί. Παράγραφος 1, ε, σημείο α, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Δέλτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Σημείο G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 4, σημείο α, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. B υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 4D υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ή e, υπέρ, κατά, δεν ψηφίζεται. Σηκώστε τα χέρια παρακαλώ. Παράγραφος 4, d υπερ κατα αποχες εγκρινεται e υπερ κατα δεν ψηφιζεται σηκωστε τα χερια παρακαλω παραγραφος 4 σημειο ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5, σημείο B, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σημείο C, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 5, σημείο ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. F, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Σημείο 5G, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 6α υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Παράγραφος 6 σημείο α, A. Ε. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Πέρας της φοφορίας. Παράγραφος 6. Έχουμε πολλές ακόμα, ε. Μην κουραζόσαστε από τώρα. Σημείο Β, Β υπέρ. Β, Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6D υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 7 D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Καλά. 7D λοιπόν. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Εγκρίθηκε. 7F υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7G υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7H υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάλι παράγραφος 8, τώρα παύλα 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παύλα 8, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παύλα 9, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παύλα 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μεγάλη γνωμοδότηση πράγματι. Παράγραφος 8 πάντα. Παύλα 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές Δεν είδα οι σοσιαλιστές. Ενρίκε υπέρ ή κατά. Υπέρ. <clears throat> Ωραία. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8, Παύλα 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παύλα 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παύλα 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παύλα 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παύλα 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παύλα 35 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παύλα 36 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παύλα 39 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9 Παύλος, Παύλα 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παύλα 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παύλα 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παύλα 8. Υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε για την Παράγραφο 9, παύλα 8. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας εγκρίθηκε. Παύλα 9. Υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε. Παύλα 9, στην παράγραφο 9. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της φοφορίας εγκρίθηκε. Τελική ε, ψηφοφορία τώρα. Ψηφίστε παρακαλώ, ηλεκτρονικά πάντα. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Με μεγάλη πλειοψηφία. Με μία αποχή. Ευχαριστούμε Μαρία Χόιμπουχ. Συγχαρητήρια για την έκθεση αυτή. Μπράβο. Και συνεχίζουμε. Και περνάμε στο σημείο 11. Ψηφίζουμε γνωμοδότηση στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς. Εδώ έχουμε πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες. Ξεκινάμε με την τροπολογία τη συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Και τώρα πάμε απευθεία στην συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχέ, έλεγχο. Για τη συμβαστική 3 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα μπορείτε να πείτε στους σοσιαλιστές ότι υπάρχει ένας παραπάνω. Ε, ο Ρίκη από τη έφυγε, αλλά είναι ένας παραπάνω. Για να βλέπω καλύτερα πώς ε, ψηφίζεται. Εάν μπορεί κάποιος να κάτσει στη σωστή θέση του σοσιαλιστές. Συμβαστική 4. Σελίδα 3 του καταλόγου. Υπέρ. Σελίδα 3 στον κατάλογο. Υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος για τη συμβαστική 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Η Έλλη θα σας δείξει πώς ψηφίσετε στους σοσιαλιστές. Εψήφισαν άπαντες. Ναι, έχετε μπερδευτεί. Ε, κρίμα. Ε, εψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνεται. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Να δείχνετε ξεκάθαρα τι ψηφίζετε γιατί τελειώς θα κάνουμε διπλό χρόνο. Ε, 21 ε, κατά τμήματα. 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεν ξέρω γιατί είναι έτσι ο κατάλογος. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πού πάμε. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε έλεγχο. Έλεγχο για το 34. 34 άρχεται η ψηφοφορία. Ευσύ ανάπαντες Πέρας. Απορρίπτεται. 36, 35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 43 υπέρ, με προφορική τροπολογία από τους πρασίνους, υπέρ, με την προφορική τροπολογία. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ήταν ενιαία ψηφοφορία για την προφορία και και τα τμήματα. Και τώρα τελική ψηφοφορία, όπω τροποποιήθηκε το κείμενο με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Όχι, μπορούμε βέβαια να το συσχυρώσουμε επειδή είναι κομμαδότηση. Όχι, όχι. Με ενδιαφέρει αν μπορώ να κάνω την ψηφοφορία τίποτα άλλο. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Να ξαναρχίσουμε μια μικρή τεχνική καθυστέρηση. Άρχεται η ψηφοφορία για το σύνολο της νομοδότησης. Ψηφίζουμε ακόμα. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, Ιγνάτσιο, για τη δουλειά σου. Σημείο 12. Θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγή για του σκοπού κοινών διαδικασιών που αφορούν τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτο διεθνού προστασία. Τα συζητήσαμε και το πρωί. Σύντομο κατάλογο, δεν θα μα πάρει πολύ. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 1. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. αποχέ Εγκρίνεται. 10. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Έλεγχο για τη 10. έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με μικρότερη διαφορά από ό,τι περίμενα. 11 τώρα. Η δύο καταπίπτει. 11 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Θα κάνουμε έναν έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τρία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τέσσερα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο σύνολο της γνωμοδότησης, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας εγκρίνεται με 14 προς 2. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Τώρα περνάμε στο 13, στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης, ανθρώπινα δικαιώματα και μετανάστευση στις τρίτες χώρες. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 8. Καταπίπτει. Κατέπεσε. Και πάμε στην 10. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. αποχέ. Έλεγχο Ελέγχουμε για τη 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. απλώ δεν είχατε συγχρονιστεί. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Δεύτερη πρόταση. Υπέρ. Κατά. εποχέ Έλεγχος. Έλεγχος για τη δεύτερη πρόταση τη 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντε πέρα Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά. Εποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Εποχές Απολύπητο. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος για την 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Σας παρακαλώ. Εάν μπορούσε ένας από την κάθε ομάδα να μας δείχνει τι ψηφίζεται, θα ήταν πολύ πιο απλό. 25, όχι 24, δεύτερη πρόταση. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28, 28 με συγχωρείτε. 28 υπέρ. Κατά. αποχέ, Αγκρίνεται. 31 υπέρ. Κατά. αποχέ. Έλεγχος. Έλεγχος για το 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα Απορρίφθηκε. Απορρίπτω το. Απορρίπτω το μια ψήφο διαφορά. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική συμβαστική 2 στην αναθεωρημένη της εκδοχή από ό,τι μου λένε. Αυτή που σας στείλαν σήμερα την ώρα της διακοπής για το γεύμα. Κυρία Γκούθμαν, για την αναθεωρημένη εκδοχή της τροπολογίας ψηφίζουμε, σωστά. Ωραία. Η αναθεωρημένη εκδοχή την έχετε δει σήμερα στο διάλειμμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το για τι ε, επιμέρου τροπολογίε. 40 υπέρ. Κατά, αποχέ. εγκρίνεται. 42 υπέρ. Όχι, δεν καταπίπτει. Όχι, όχι, όχι, γιατί η συμβαστική δεν έγινε δεκτή. 42. Είναι ασύμβατη. Όχι, όχι, όχι. Η συμβαστική ε, απορρίφθηκε. Η 40 έγινε δεκτή, η 42 είναι ασύμβατη με τη 40. Αυτό είναι το ερώτημα. Μισό λεπτό να το ελέγξουμε. Yes, I I mean... Ναι, ναι, κατάλαβα, αλλά μου λένε ότι είναι ασύμβατη η 42. Θα έπρεπε να καταπέσει. Επειδή γκρίναμε την 40, να ψηφίσουμε τη 42, τι λέτε εσείς. Ε, μπορεί απλώς να απορριφθεί. Είναι πιο απλό. Να την ψηφίσουμε και αν δεν θέλετε να το απορρίψουμε. Είναι πιο εύκολο από το να ελέγξουμε. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, συγγνώμη, 40 έγινε. 42. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Λοιπόν, και τώρα το σύνολο της νομοδότησης διαλεκτρονικής ψηφοφορίας άρχεται. Εψήφισαν άπαντας. Πέρας. Γίνεται δεκτή 20 προς 2. Ευχαριστούμε την εισηγήτρια την κυρία Κούφμαν. Σημαντική έκθεση του κυρίου Νταν Πρέντα για την αναπτυξιακή πολιτική και τη συνοχή της. Έκθεση Νταν Πρέντα σημαντική έκθεση. οι συζητήσεις εκτός αιθούσης. Σημαντική έκθεση για την συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη μου χαρά να μπορώ να ευχαριστήσω τις άλλες πολιτικές ομάδες. Σας παρακαλώ, έχει πηγαδάκια μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης τα πηγαδάκια σας εκτός. Κύριε Πρέντα, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφου από τι άλλες πολιτικές ομάδες για τη συνεργασία μας. Ελπίζω ότι θα συνεχιστεί ε, ψηφίζοντας κατά του ΕΛΚ σήμερα. Okay, we, we start the vote. Λοιπόν, αρχίζουμε την ψηφοφορία. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Η συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ, κατά αποχές δεκτή νομίζω έλεγχος έλεγχος 34 άρχεται η ψηφοφορία ε, ψήφισαν όλοι πέρας δεκτή με διαφορά μιας ψήφου πολύ κοντά συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 κατά 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 44 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή Ε, συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τμηματική στη 49. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 58 υπέρ κατά αποχές έλεγχος έλεγχος την 58 την 58 άρχεται όχι ναι 58 άρχεται ψηφοφορία πέρας δεκτή συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές δεκτή 68 ε, υπέρ κατά αποχές έλεγχος έλεγχος είναι 68 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή μια ψήφο διαφορά τμηματική στην 69 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές δεκτό Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Το δεύτερο τμήμα άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Κατα... Η 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 73, α, τμήματική. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Έλεγχος. Το πρώτο του 70 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτό. Δεύτερο τμήμα της 73. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, κάναμε και στο 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Το δεύτερο τμήμα ηλεκτρονικά το ψηφίζουμε. Πέρας. Δεκτό. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχο στην 74 δεν βλέπω. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή. Τμήματική στην 75 πρώτο τμήμα. Υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. Υπέρ κατά αποχές δεκτό. 78 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Την 78. Άρχεται η ψηφοφορία για την 78. Πέρας. Δεκτή. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 88 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 93 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Α, έλεγχο αν θέλετε να... Ε, δεκτή. Ε, υπέρ, κατά, εποχές. 100 in favor. 100 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρι... Να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Απορρίπτεται. 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 105. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 105. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε έλεγχο για την 106. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική 16. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη. 114 υπέρ κατά έλεγχος. Ελέγχουμε για την 114. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ξεχωριστή, σε, κατά ψηφοφορία για την 122. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Έλεγχος για το πρώτο τμήμα της 122. Άρχεται η ψηφοφορία. Με ψήφισαν άπαντε. Πέρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 124. 124 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 140 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στις αναφορέ. αναφορές. Ετελογική αναφορά 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά τροπολογία 2 εγκρίνεται. 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος, έλεγχος για την 5. Άρχεται η ψηφοφορία. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Μία ψήφος διαφορά. Δίκαιο. Είχατε πολύ κοντά. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Έλεγχος για την ψηφοφορία, για την τροπολογία, συγγνώμη, 6. Εψήφισαν άπαντες. Πέρας. Εγκρίνεται. Επτά. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γνωμοδότηση ίντα. Μπορούμε να τα ψηφίσουμε unblock όλα μαζί. Θα τα ψηφίσουμε on block. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι τροπολογίες ήρθα εγκρίνονται. Οπότε τώρα ψηφίζουμε ηλεκτρονικός συνολικά την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία συνάδελφοι. Εψήφισαν άπαντες πέρας. Κύριε Πρέντα, έχετε πολύ μεγάλη πλειοψηφία με δύο αποχέ μόνο. Μπράβο σας. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να φύγετε ησύχω διότι θέλω να περάσουμε πολύ γρήγορα στο σημείο 15. 15 προετοιμασία τη μετακλογική αναθεώρησης του ΠΟΥΔΟΠΟΥ. Ο συγκεκριτής μας είναι ο κύριος Ρούμπιχ, του δίνω το λόγο και παρακαλώ να φύγετε ήσυχο. Κύριε Ρούμπιχ. Sorry, Rubik, we're moving to item 15. Sorry, can people leave quietly? Να αποχωρήσετε ησύχω, παρακαλώ. Όλοι. Κύριε Ρούμπικ, το 15. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η ενδιάμεση αξιολόγηση είναι για μας μεγάλη πρόκληση. Είδαμε ότι τα τελευταία χρόνια σε αυτό το τομέα έχουν αλλάξει πολλά και γι' αυτό η ευελιξία και οι απαιτήσει και οι νέε προκλήσεις πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης. Ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες είδαμε ότι ο κόσμος δεν είναι πια διατεθειμένος να παραμείνει αλλά όλοι επιθυμούν να φτάσουν στη, στη σταθερή Ευρώπη. Δεν θέλουμε να γνωρίσουν την αρχή η φτώχεια για όλους λίγοι μόνο, 0,00% ε, πλουτίζουν και μάλιστα με, με πάνω στη βάση της διαφθοράς δεν μπορεί να εφαρμοστεί η κοινωνική οικονομία της αγοράς σε αυτές τις χώρες. Και το ερώτημα που τίθεται για όλους εμάς είναι αν η αναπτυξιακή πολιτική όπως την ασκούσαμε μέχρι τώρα και στα πλαίσια της οποίας πολλά χρήματα ε, δαπανούνταν, όπως και ιδεαλιστικές στρατηγικές, αν αυτή η αναπτυξιακή πολιτική στέφθηκε από επιτυχία ή μήπως πρέπει να ξαναγυρίσουμε στα βασικά της ανάπτυξης και ποια είναι τα βασικά. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις που διασφάλιζαν την ευημερία σε μια κοινωνία. Ίσως λοιπόν στο μέλλον πάλι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτή την πολιτική. Τότε οι γυναίκες ήταν υπεύθυνε για την οικογένεια αλλά και για την επιχείρηση πολλές φορές. Ίσως λοιπόν θα πρέπει η οικογένεια να τεθεί στο επίκεντρο και η μεικτή οικονομία θα πρέπει να συνοδεύεται από εμά και από τεχνική βοήθεια και υποστήριξη για να μπορέσει ο στόχος βιώσιμης ανάπτυξης 16 για την ειρήνη, ασφάλεια και δικαιοσύνη να τεθεί στο επίκεντρο. Η ευημερία αρχίζει όταν υπάρχουν ενεργειακοί πόροι. Χωρίς ενέργεια δεν μπορεί κανείς να συνδεθεί με τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας δεν έχει φως για να δουλεύει, δεν μπορεί να φροντίσει για την ασφάλεια. Και έτσι η ενέργεια πιστεύω ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα ιδιαίτερα στην Ήπεθρο, ούτω ώστε να εξασφαλιστούν συνθήκες εργασίας και προϋποθέσεις για τον πληθυσμό που θα μπορέσουν να οδηγήσουν σε ευημερία και ανάπτυξη. Συμφωνούμε ότι οι χώρες, τις λιγότερο αναπτυγμένες ε, χώρες, ε, πρέπει να βοηθηθούν αλλά αυτό θα γίνει μέσα από επενδύσεις. Επενδύσεις στην παιδεία, στην μετεκπαίδευση, την επιμόρφωση, στην διαδική ε, επαγγελματική κατάρτιση, ε, επενδύσεις σε δομές, ε, που θα ενισχύσουν τη δικαιοσύνη, τις εισαγγελίες, ε, φροντίζοντας ε, για διαφάνεια και σωστό καταμερισμό και διάκριση των εξουσιών. Η διάκριση των εξουσιών και η οικολογική και κοινωνική οικονομία της αγοράς είναι προτεραιότητες. Το 0,7% του ακαθάριστου εγχώριου εισοδήματος θα πρέπει να το διαθέσουμε. Επίσης, η διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή ε, έδειξε κάποια συμπεράσματα ε, που αφορούν τις εκπομπές και την λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Καλό είναι λοιπόν να ληφθούν υπόψη όπως και οι ε, προσπάθειες για καθαρό νερό, ε, ατμόσφαιρα ε, και πρώτες ύλες. Αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην ενδιάμεση αξιολόγηση. Στην πραγματικότητα, οι στόχοι της Ένωσης στην ενδιάμεση αξιολόγηση θα πρέπει να εναρμονιστούν με τους στόχους της αναπτυσσόμενες χώρες και να ε, υποβοηθηθούν να αναβαθμίσουν τα πρότυπά τους. Αυτά τα θέματα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων. Ε, κάνω έκκληση στους Υπουργούς Οικονομικών των κρατών μελών να μην ε, επιμείνουν στις ε, ε μειώσεις. Αντιμετωπίζουμε μεγάλη πρόκληση και αυτή θα αντιμετωπιστεί με θάρρος, με ε, δέσμευση από την πλευρά μας. Γι' αυτό η Επιτροπή μας είναι πολύ σημαντική από αυτή την άποψη, διότι θα πρέπει να ε, αναθεωρήσουμε αυτά που ήταν λιγότερο αποτελεσματικά ε, από αυτά που κάναμε να δούμε τι, ήταν, τι δεν ήταν αποτελεσματικό και να το αλλάξουμε ε, σε συνδυασμό και με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις ε, που δικούνται από γυναίκες, οι ε, οικογενειακές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο. Αυτό το θεματολόγιο δεν ισχύει μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά περισσότερο για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης οι νέοι επιχειρηματίες θα πρέπει να υποστηριχθούν, να βοηθηθούν και επιτόπου εδώ ερχόμενοι στην Ευρώπη μπορούν να μάθουν πώς θα δημιουργήσουν υποδομές και σε τελευταία ανάλυση πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα των καινοτομιών. Μετά θα ε, εφαρμόσουν με προσαρμογές βέβαια τα όσα έμαθαν στη χώρα τους. Αυτή η ε, στόχη του πολιετούς προγράμματος 14-20 ε, θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Νομίζω ότι όλες οι πολιτικές ομάδες ε, συμφωνούν ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και να φροντίσουμε για ένα επίπεδο ευημερίας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και δεν γίνεται αυτό μόνο με αναδιανομή, αλλά και με εργασία, εξειδικευμένη εργασία, με επιμόρφωση και μετεκπαίδευση. Ευχαριστώ. Καλώ συνάδελφοι. Τώρα έχουμε εδώ τον προσκεκλημένο μας από το λεκτικό συνέδριο. Όταν έχουμε τις τροπολογίες να συζητήσουμε με τους χιώδεις, αν συμφωνείτε, τι λέτε, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν έχει ζητήσει το λόγο, νομίζω ότι αυτό θα ήταν καλύτερα να κάνουμε για να ακούσουμε το λεκτικό συνέδριο. Έτσι καλώς έχει να κάνει και με αυτό που είπατε εσείς. Να δούμε τελικά που ακριβώς θα είναι η προτεραιότητά μας. Εντάξει, δεν θα συζητήσουμε τώρα, συνάδελφοι. Θα συζητήσουμε όταν έχουμε τις τροπολογίες. Η προθεσμία είναι Απριλίου και θα ψηφίσουμε στις 24 Μαΐου. Λοιπόν, Αφήνουμε λοιπόν το σημείο αυτό, το 15, στην ημερήσια διάταξη και συνεχίζουμε. Okay, sorry, I'm looking at the number there. I will move, leave item 15 and move now to item 16. And I'm therefore very, very pleased to meet Mr. to welcome Mr. Pinkston. Καλωσορίζω τον κύριο Πίξεν εδώ και τον κύριο Λένε. που θα μας μιλήσουν. Ναι, πριν ε, να είμαι εγώ εδώ. Δεν το ήξερα. Θα μας πείτε πότε ήσασταν στο Κοινοβούλιο σε λίγο. Λοιπόν, προχωράμε στο σημείο 16 και για τη σημερινή συζήτηση έχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, η Επιτροπή μας παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων για την αναπτυξιακή βοήθεια. Κάθε χρόνο έχουμε έκθεση για την απαλλαγή, για το πώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια. Κατά το παρελθόν δεν είχαμε τόσο σε βάθος συζήτηση για το τι πρέπει να κάνουμε. Οι συντονιστές αποφάσισαν να έρθει το ελεγκτικό συνέδριο εδώ και να συζητήσουμε μαζί σε βάθος. Πρώτα θα ακούσουμε τον Κάρελ Πίνγκστεν, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος θα μιλήσει γενικώ για την αναπτυξιακή βοήθεια και πώς ε, ελέγχεται αυτή. Και στη συνέχεια θα μας πείτε πώς πιστεύετε ότι μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να βελτιώσει το δικό του έλεγχο. Όταν θα έχουμε τελειώσει λοιπόν με τον κύριο Πίνξτεν, τότε θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Λένε, που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, που είναι υπεύθυνο για την ε, διευκόλυνση, την επενδυτική διευκόλυνση. Λοιπόν, κύριε Πίνξτεν, έχετε το λόγο. Να μας πείτε και πότε ήσασταν εδώ στο Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μας καλέσατε. Έχουμε και τον κύριο Φαντζίου μαζί μας, το διευθυντή μας. Καλό είναι να τον γνωρίσετε. Είναι διευθυντής του Σώματος 3 που ασχολείται με τις εξωτερικές δράσεις. Για σηκωθείτε να σας δουν όλοι ποιος είσαστε. Να, αυτός είναι. Ναι, ήμουν ευρωβουλευτή. Για να απαντήσω στην ερώτησή σας, για λίγο βέβαια, ένα σύντομο χρονικό διάστημα, στο τέλος της προηγούμενης χιλιετία, το 89 εξελέγει, και μετά ασχολήθηκα με την εθνική πολιτική που βρήκα, με απόλυτη ειλικρίνεια το λέω, λιγότερο ενδιαφέρουσα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά δεν αποφασίζει κανείς πάντα από μόνος του τι θα κάνει και ποιες είναι οι προοπτικές. Έτσι έχουν τα πράγματα στην πολιτική. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μας καλέσατε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και θα σας κάνω μια γενική εισαγωγή. Ξέρω ότι οι ευρωβουλευτές εδώ δεν είναι πάντα εξίσου εξοικειωμένοι όπως και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμών στους οποίους παρουσίασα τα θέματα αυτά το πρωί. Λοιπόν, το ελεκτικό συνέδριο, όπως γνωρίζετε, είναι ένα θεσμικό όργανο, προβλέπεται από την συνθήκη και είναι το ελεγκτικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ως ελεγκτής προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι για τους εταίρους μας και ένας από αυτούς είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι Ευρωβουλευτές, αλλά και το Συμβούλιο φυσικά, και βέβαια οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι γενικότερα. Ό,τι εκθέσεις ε, ετοιμάζουμε, οι αιτήσει εκθέσεις μας για παράδειγμα, χρησιμεύουν στη διαδικασία απαλλαγής. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να σας πω. Τώρα, πιο συγκεκριμένα για το σώμα 3 του ελεκτικού συνεδρίου. Έχουμε αυτό που λέμε τα κάθετα σώματα. Ένα είναι για την γεωργία, το σώμα 3 είναι αυτό το οποίο ασχολείται με τις εξωτερικές μας δράσεις. Αυτό σημαίνει ότι ελέγχουμε τις δαπάνες κονδυλίων που πάνε στην εξωτερική μας πολιτική. Ελέγχουμε τις δαπάνες για τις υποψήφιες χώρες και τις ενδυνάμει υποψήφιες χώρες και ελέγχουμε και την αναπτυξιακή βοήθεια και την ανθρωπιστική βοήθεια που δίνεται στις αναπτυσσόμενες αλλά και στις γείτονες χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός, ξέρετε, ποιος είναι, 65 δις για την περίοδο τώρα την τελευταία μέχρι το 2020. Πώς γίνεται αυτό. Βασικό είναι να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τριών ειδών έλεγχοι. Όταν μιλάμε για χρηματοδοτικό έλεγχο, δημοσιονομικό έλεγχο, αυτό σημαίνει ότι εξετάζουμε την εξοπιστία των λογαριασμών, κατά πόσο οι λογαριασμοί δηλαδή αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Όταν μιλάμε για συμμόρφωση, μιλάμε για συμμόρφωση με την ομοθεσία, με τους κανονισμούς, με τις ρυθμίσεις που ισχύουν. Κοιτάμε δηλαδή και την νομιμότητα και την κανονικότητα και στη συνέχεια έχουμε και τις επιδόσεις, τον έλεγχο επιδόσεων, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για σας. Όταν μιλάμε για έλεγχο των επιδόσεων, σημαίνει ότι κοιτάμε κατά πόσο ορθά έγινε η διαχείριση των ε, κονδυλίων. Αν πιάσαν τα λεφτά μας τόπο, με δύο λόγια. Οπότε θα μπω τώρα στην ουσία και στις λεπτομέρειες αυτού του τρίτου σκέλους, της επίδοσης. Σχεδόν πάντα πρόκειται για το αν πιάνουν τόπο τα λεφτά μας, ποιες είναι οι επιδόσεις μας. Στις ειδικέ μας εκθέσεις προσπαθούμε να δίνουμε στοιχεία κάθε φορά που υπάρχει ανεπαρκής επίδοση στους ελέγχους που κάνει το ηλεκτρικό συνέδριο αν δεν υπάρχουν νέα, αυτό είναι καλό νέα. No news, good news. Δεν είμαστε όπως οι δημοσιογράφοι εμείς, δεν θέλουμε νέα, προτιμάμε να μην έχουμε. Που σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Συνήθως εντοπίζουμε τα αρνητικά. Επού και πού λέμε και κάτι ιδιαίτερα θετικό αν έχουμε διαπιστώσει κάτι εξαιρετικό από πλευρά τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις δικές μας λοιπόν εκθέσεις αναφέρουμε κυρίως αυτό που στα αγγλικά είναι τα τρία E, δηλαδή είναι effectiveness, η αποτελεσματικότητα, που σημαίνει ότι κοιτάμε κατά πόσο οι προθέσεις υλοποιήθηκαν. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από τα τρία ε, στα αγγλικά τουλάχιστον. Το δεύτερο έχει να κάνει με την απόδοση, με την σχέση δηλαδή της προσπάθειας που έχει γίνει της οικονομικής με τα αποτελέσματα. Και στη συνέχεια έχουμε και την οικονομία, δηλαδή αν δεν έχουν σπαταληθεί χρήματα. Αυτό προσπαθούμε να βρούμε. Ότι δηλαδή τα κονδύλια δαπανήθηκαν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Economy, efficiency και effectiveness είναι τα τρία ε στα αγγλικά. Συνήθως με την αποτελεσματικότητα λοιπόν ασχολούμεθα. Στο δικό μας σώμα, το σώμα 3 όπως είπαμε, έχουμε κατά μέσο όρο 6 ειδικέ εκθέσεις ετησίως. Και αν δείτε τους πόρους που διαθέτουμε, θα έλεγα ότι είμαστε το πιο παραγωγικό σώμα του ελεγκτικού συνεδρίου με τόσες πολλές εκθέσεις. Και αυτό οφείλεται όχι μόνο στα μέλη μας, αλλά και στο προσωπικό μας, το οποίο δουλεύει σκληρά. Θα σας δώσω τώρα μερικά παραδείγματα για τις επιδόσεις μας από το 2015. Το πρώτο παράδειγμα είναι η αποστολή τη UPOL στο Αφγανιστάν. Τι βρήκαμε εκεί, τι διαπιστώσαμε. Επρόκειτο για την μεταρρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών στο Αφγανιστάν και για την επαγγελματική διάσταση της αστυνομίας. Και το συμπέρασμά μας είναι ότι η διαχείριση ήταν ικανοποιητική από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειώσαμε κάποια αρνητικά, αλλά γενικά ήταν θετικό. Το δεύτερο ήταν η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση των βασανιστήριων. Ο κύριος Λένε θα σας πει περισσότερα γι' αυτό. Εδώ καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή δεν, έβαλε, δεν έλαβε υπόψη τις επαρκώς τις προτεραιότητες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, στις διάφορες χώρες που εξέτασε. Πολλά θα μπορούσε κανείς να προσθέσει εδώ. Και η άλλη παρατήρησή μας ήταν για την έλλειψη συντονισμού με άλλες δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τρίτο παράδειγμα. Πάλι από το 2015 η έκθεση για τις χώρες που παράγουν κασίταρο, το πρόγραμμα δράσης. Και εδώ είπαμε ότι η Ευρωπαϊκή... Συγγνώμη, για ξυλία πρόκειται. Και εδώ είπαμε ότι τα κύρια προγράμματα που εξετάσαμε δεν ήταν επιτυχή και ότι οι αδειοδοτήσεις και τα προγράμματα αδειοδοτήσεων δεν λειτουργούσαν πλήρως σε καμία από τις χώρες ε, εταίρους. Σε καμία. Κάτι άλλο τώρα. Ενεργειακή απόδοση στην Ανατολική Αφρική. Εδώ σημειώνεται κάποια πρόοδος, κάποια επιτυχία και συμπεράναμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε καλή επιλογή μεταξύ των προγραμμάτων που προτάθηκαν, αλλά υπήρχαν κάποια προβλήματα και αποτυχίες στον έλεγχο υλοποίηση των προγραμμάτων. Και κάτι άλλο είναι το θέμα για το οποίο θα σας μιλήσει ο κύριος Λένε, που είναι δηλαδή η επενδυτική διευκόλυνση. Μια δική έκθεση δεν είχε να κάνει με δαπάνες, γιατί περιμένετε ότι τι ελέγχουμε, ελέγχουμε τις δαπάνες. Ε, λοιπόν, σήμερα το πρωί την παρουσίασα στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών είχε έναν περίπλοκο τίτλο. Πρόκειται για αναθεώρηση των κινδύνων όσον αφορά τις αναπτυξιακές δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν νομίζω πολύ χρήσιμο τα μέλη της Επιτροπής σας να ενημερωθούν για την έκθεση αυτή και θα μπορούσατε να ζητήσετε από το προσωπικό επίσης να ενημερωθεί. Είναι κάτι που παρουσιάσαμε στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμών. Η προσέγγισή μας, λοιπόν όσον αφορά τα αποτελέσματα, είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει μόνο το τι δαπανάτε, αλλά και τα αποτελέσματα των δαπανών αυτών. όταν κάποιος έχει έναν προπολογισμό, είτε πρόκειται στο ιδιωτικό τομέα είτε στο δημόσιο, φροντίζει και προγραμματίζει τις δαπάνες να γίνουν μέσα στη χρονιά. Έχουμε εντοπίσει εννέα περιοχές κινδύνου όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. λέμε ότι οι στόχοι πρέπει να είναι ευφύς. Smart. Αλλά βέβαια το smart είναι ακρονίμιο. Έχει να κάνει με δίχτες μερικές φορές, ενώ πρέπει να έχει να κάνει με στόχους. Οι δείκτες λέμε πρέπει να είναι σαφείς και είναι κάτι το οποίο διαφοροποιείται από τους στόχους. Άλλο δείκτες, άλλο οι στόχοι. Εδώ δεν πρόκειται για χρήματα δηλαδή, αλλά πρόκειται για κινδύνους που ελοχεύουν στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ άλλων για την και βοήθεια. Πριν ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου να σας πω ότι μερικές φορές υπάρχουν επικρίσεις επειδή μας λένε ότι οι αιτήσεις εκθέσεις μας είναι πολύ τεχνικές. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι όταν διαβάζει κανείς μία ειδική έκθεση ή ένα κεφάλαιο από έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, φυσικά δεν είναι σαν να διαβάζει εφημερίδα. Είναι πιο εύκολο μερικές φορές να διαβάζει κανείς ακόμα και τους Financial Times ή τη Mondi ή την El País από το να διαβάζει τις δικές μας ειδικέ εκθέσεις. Δεν είμαστε όμως δημοσιογράφοι, συνεπώς πρέπει να ακολουθούμε απολύτως τους κανόνες και τους τύπους όπως πρέπει να τα κάνουμε, έτσι να τα κάνουμε. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε γλώσσα κατανοητή και καμιά φορά λέμε ο ένας τον άλλον ξέρεις τα κείμενά μας πρέπει να διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο που να τα καταλαβαίνει ο καθένας. Εντάξει, δεν λέω ότι οι ευρωβουλευτές είναι ο καθένας. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε σαφή διατύπωση. Και τέλος και θα δώσω το λόγο στον κύριο Λένη, εσείς θα το δώσετε τέλος πάντων, κάποιοι πιστεύουν ακόμα και το Κοινοβούλιο ότι όταν επιλέγουμε τα καθήκοντά μας είναι σαν να το ρίχνουμε στα ζάρια. Ε, όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η επιλογή των αρμοδιοτήτων μας, των καθηκόντων μας, είναι κάτι που γίνεται με πολύ ρυθμισμένο τρόπο. Έχουμε καταρχήν την έγκριση του ετησίου προγράμματός μας. Βάσει κριτηρίων. Και ποια είναι αυτά. Πρώτα απ' όλα το συμφέρον των ενδιαφερόμενων πλευρών και ελέγχουν το προσωπικό μας δηλαδή όλα τα έγγραφα που έχουμε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Απαλλαγές, οτιδήποτε. Όλα αυτά τα εξετάζει το προσωπικό μας. Οπότε αν κάτι δεν κολλάει καλά, λέμε α, πρέπει να ελέγξουμε και τα υπόλοιπα κριτήρια. Κοιτάμε το επίπεδο κινδύνου. Δεν έχει νόημα να πανάμε από πριν αν ξέρουμε ότι με τον έλεγχο θα αποδειχτεί ότι δεν υπάρχει ίχνος κινδύνου. Είναι χάσιμο χρόνο και χρήματος. Κατάχρηση πόρων, αν υπάρχει μηδαμινός κίνδυνος και κοιτάμε και την δυνάμει προστιθέμενη αξία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα τέτοια προστιθέμενης αξίας. Παράδειγμα, πέρυσι είχαμε μια ειδική έκθεση για τη u στο Αφγανιστάν, όπως σας είπα. Δεν έχει νόημα να ξανακάνουμε το ίδιο την επόμενη χρονιά. Το κάναμε πέρυσι. Δεν το ξανακάνουμε και φέτος. Δεν θα υπήρχε προστιθέμενη αξία αν το ξανακάναμε φέτος. Οπότε κοιτάμε ποια θέματα, ποιες χώρες έχουν καλυφθεί τα πρόσφατα έτη και δεν το επαναλαμβάνουμε. Είναι και αυτό ένα κριτήριο δηλαδή. Μπορώ επίσης να σας πω ότι χτες στη συνεδρίαση που είχε το Σώμα 3 αποφασίσαμε για έλεγχο όσον αφορά την προσφυγική κρίση και επικεντρωνόμαστε στα hot spots. Καταλαβαίνετε ότι είναι κινούμενο στόχος για μα. έτσι. Αλλά θέλουμε να προσπαθήσουμε να τελειώσουμε μέχρι τα τέλη της χρονιάς, γιατί αλλιώ δεν θα έχει νόημα. Είναι βάση συγκεκριμένων κριτηρίων και στόχων το άργο μας, το ελεγκτικό. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για την υπομονή σας, για την προσοχή σας και εκ μέρου των συναδέρφων από το Σώμα 3 μπορώ να σας πω ότι θα συνεχίσουμε να σας βοηθούμε, να σας ενημερώνουμε, να σας πληροφορούμε για τα τεκτενόμενα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. I think um, said Ευχαριστώ πολύ. Μας είπατε πολλά και σημαντικά. Δουλεύετε πάνω σε θέματα που όντως και μας μας ενδιαφέρουν πολύ. Το συζητήσαμε και το πρωί για το προσφυγικό, για παράδειγμα. Τώρα στο Κοινοβούλιο συχνά έχουμε την αίσθηση ότι εσείς δουλεύετε πάνω στα νούμερα, ότι προσθέτετε, αφαιρείτε και δεν είναι αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς. Όντως πιο πολύ μας ενδιαφέρουν οι επιδόσεις, η απόδοση κλπ. Κάτι άλλο σημαντικό που μας είπατε είναι ότι ερευνάτε προγράμματα στο οποίο λοχεύει κάποιος κίνδυνος. Εμείς λέμε ότι κάθε φορά που λέει το Λεκτικό συνέδριο ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, αυτό είναι αρνητικό. Μα έτσι κι αλλιώς η ανάπτυξη γίνεται σε έναν χώρο που ελοχεύει κίνδυνος. Δεν θα μπορούσαμε να λειτουργούμε μόνο ελήψη κινδύνου, δεν θα έχει δουλειά και το Λεκτικό συνέδριο τότε. Είναι λογικό η αναπτυξιακή βοήθεια να συνδέεται με τον κίνδυνο. Πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι συνάδελφοι. Δεν σημαίνει κάθε φορά που εσείς εντοπίζετε κάποιο πρόβλημα και εκφράζετε κριτική ότι πρέπει να σταματήσουν και τα σχετικά προγράμματα. Λοιπόν, κύριε Λένε, εσείς τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ χαίρομαι που επιστρέφω στο Κοινοβούλιο σήμερα για να παρουσιάσω ε, ένα θέμα στην Επιτροπή Ανάπτυξης που είναι ο πρώτος. Ε, βέβαια, η, ε, συνήθως ε, οι νομοθετικά υπεύθυνε επιτροπές είναι οι επιτροπές οι άλλες εκτός από την Επιτροπή Προϋπολογισμών που παρουσιάζουμε εμείς τα θέματά μας. Τι επενδυτική διευκόλυνση είναι αυτή. Είναι ένα ταμείο το οποίο αποτελείται από κονδύλια των κρατών μελών και της, της Τράπεζας Επενδύσεων ήταν περίπου 4,5 δις ευρώ τα προηγούμενα 10 ε, χρόνια. Εμείς έχουμε περιορισμένες δυνατότητες ελέγχου και βάσει της οργανικής Συμφωνίας μεταξύ του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό είναι ένα ανανεώσιμο ε, κεφάλαιο, ε, ε, οικονομικά δηλαδή είναι βιώσιμο και αηφόρο. Ε, πάνω από 5 δις ευρώ τα προηγούμενα 10 χρόνια χρησιμοποιήθηκαν για αναπτυξιακά προγράμματα. Η διευκόλυνση επικεντρώνεται σε επιστοτικές γραμμές για χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, κεφάλαιο κινδύνου, χρηματοδότηση έργων υποδομής είναι δηλαδή ε, ιδιωτικά έργα τα οποία έχουν ε, δημόσια σημασία. Αυτός είναι ο στόχος. Εμείς κάναμε τον έλεγχο γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας παρακάλεσε, μας εκάλεσε να ε, κάνουμε μια έκθεση. 20 ήταν τα έργα που ελέγχθηκαν, 35% ε, υπογεγραμμένες συμβάσεις από το 2011 μέχρι το 2014 και διάφορα χρηματοδοτικά μέσα και οικονομικοί τομείς ε, καλύφθηκαν από εκεί. Ε, ε αυτά, ο έλεγχος έγινε στα πλαίσια ε, γρήγορων ειδικών εκθέσεων ε, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο του 2015. Τότε, σε αυτό το διάστημα, καταρτίστηκε η έκθεση. Ε, εδώ έχουμε ένα νέο μέσον το οποίο έχει ε, προσθεθεί και έχουμε και το πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ήταν το πρώτο ούτω ώστε γρήγορα να ανταποκρινόμεθα ε, στις απαιτήσει των εμπλεκομένων. Καταρχήν, ε, εμείς ε, ε, θέλαμε να δούμε δύο θέματα, δηλαδή η προώθηση από τη διευκόλυνση αυτή ε, είναι συνεπής με το, αναπτυξιακό έργο της Ένωσης. Ε, διευκολύνει ως καταλήτης μέσα από δάνεια σε τοπικό νόμισμα ούτως ώστε να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτά απαντήθηκαν θετικά. Εμείς διαπιστώσαμε ότι η χρηματοδότηση μέσω της διευκόλυνσης είναι ε, συνάδει με τη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Η Τράπεζα Επενδύσεων δεν χρηματοδοτεί τις ΜΜΕ έμεσα, αλλά μέσω πιστοτικών γραμμών προς χρηματοπιστωτικούς ε, διαμεσολαβητές. Στα πλαίσια μιας ειδική διαδικασίας κατανομής, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να διασφαλίζει ότι οι πιστώσεις φάνουν στους τελικούς δικαιούχους που πρέπει να προωθηθούν. Η Συμφωνία του Κοτονού επιτρέπει και συμμετοχές ιδίων κεφαλαίων ε, για να ε, διατεθούν σε ΜΜΕ. Αυτό γίνεται άμεσα μέσα από συμμετοχή των επιχειρήσεων ή έμεσα μέσα από ιδιωτικά equity funds. Μέσα από τις συμμετοχές ιδίων κεφαλαίων μπορεί να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, και αυτό μπορεί να είναι και μπορεί να υπάρχει και συμβολή στην ενίσχυση της ε, χρηματοπιστωτικής αγοράς της χώρας. Διαπιστώνουμε επίσης ότι οι άμεσες επενδύσεις συμφωνούν με τους αναπτυξιακούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δημιουργούν ε, προστιθέμενη αξία, την οποία εξετάσαμε μέσα από πάνω σε τρεις βάσεις. Πρώτον, οι πιστοτικές γραμμές της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, ε, επιτρέπουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί και με τοπικά νομίσματα, αναλαμβάνει έτσι το συναλλαγματικό κίνδυνο και σταθεροποιεί έτσι και τη χορήγηση των δανείων. Η Ευρωπαϊκή ε, Τράπεζα Επενδύσεων ε, πολλές φορές ε, έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε, αυτή τη, αυτό το τομέα της χρηματοδότησης με εθνικό νόμισμα. Στην Γκάνα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν δεν υπήρχε αυτό το σύστημα, η επιβάρυνση μέσα από τα επιτόκια θα ήταν τόσο υψηλή, ώστε δεν θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν τα χρήματα για την αποπληρωμή των δανείων η, επειδή διαθέτησε εθνικό νόμισμα η τράπεζα τα, τα δάνεια και με ευνοϊκούς όρους ε, μπόρεσε να μειώσει ε, το κόστος και έτσι μπόρεσαν ε, οι επενδύσεις να γίνουν, για παράδειγμα, στο αεροδρόμιο του Έντεμπε. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για το πώς ε, η ανάληψη του συναλλαγματικού κινδύνου μέσα από χρηματο πετράπη ε, μέσα από τη χρηματοδότηση σε τοπικό νόμισμα. Ε, επίσης είδαμε ότι υπάρχει μόχλευση ε, ικανοποιητική. Με τη χρηματοδότηση από την Τράπεζα Επενδύσεων, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ε, ήταν δυνατόν να προσελκυστούν και άλλοι χρηματοδότες. Ε, με το Quick Special Audit ε, δεν ε, μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία για να υπολογίσουμε ακριβώς τις, πώς θα ήταν οι επενδύσεις χωρίς την ε, συμμετοχή της Τράπεζας Επενδύσεων. δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό στα πλαίσια της ε, σύντομης έκθεσης που καταρτήσαμε. τώρα, σε ό,τι αφορά τις συστάσεις, ε, ε, λίγα πράγματα ε, μπορέσαμε να συστήσουμε γιατί ήταν θετικά τα αποτελέσματα, ο έλεγχος ήταν θετικός. Το ελεγκτικό συνέδριο έκανε δύο συστάσεις σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση πιστοτικών γραμμών που γίνονται δεκτές από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πρέπει να γίνουν δεκτές. Ένα θέμα είναι η διαφάνεια, δηλαδή ο τελικός δικαιούχος θα πρέπει να γνωρίζει ότι παίρνει χρήματα από την επενδυτική διευκόλυνση. Ο τελικός δικαιούχος πολλές φορές δεν εγνώριζε δηλαδή ότι τα χρήματα προέρχονταν από τη διευκόλυνση και από την Τράπεζα Επενδύσεων. Δεν του είχαν δοθεί ε, οι πληροφορίες. Ε, ε, ήταν παραβλεψή, αλλά αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Ε, επίσης, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να αξιοποιήσουν περισσότερο από ό,τι μέχρι τώρα την τεχνική βοήθεια και αυτό πώς θα εξασφαλιστεί αν ενημερώνονται για τη δυνατότητα που, υπάρχει για τη χρήση των χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών. Ε, αυτό είναι ένα σημείο που νομίζω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί. Δηλαδή ε, να ε, προσφέρεται και η δυνατότητα αυτή στον τελικό δικαιούχο. να γνωρίζει ότι υπάρχει και η δυνατότητα του διαμεσολαβητή. Αυτό ήταν κάτι που το παρατηρήσαμε και γι' αυτό και η σύσταση. Γενικά η συνολική μας εντύπωση ήταν πολύ καλή, εκτός από τα μικρολαθάκια που είδαμε ε, και από την East African Development Bank και οι ειδικοί του, της Τράπεζας Επενδύσεων συνεργάστηκαν πολύ επαγγελματικά και αποτελεσματικά Πήγαμε και επισκεφθήκαμε και κάποια έργα και έχουμε την εντύπωση ότι πρόκειται για πάρα πολύ αξιέπαινα εκ των προτέρων ε, ε, ε, ε ελεγμένα έργα με σημαντικό αντίκτυπο. Νομίζω ότι ε, αυτή την παρουσίαση την έκανα και στην Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών ε, και μετά απαντήσαμε σε ερωτήσεις, όπως βέβαια είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε και τώρα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Έχουμε στους φακέλους σας, συνάδελφοι, όλο τον κατάλογο με τα έργα και την παρουσίασή σας. Ευχαριστούμε πολύ για τις ομολίες σας. Έχουμε συζητήσει κάποια από τα έργα αυτά κατά καιρού και ήταν σημαντικό να ακούσουμε και τη δική σα οπτική γωνία. Έχω πολλούς ε, εισηγητέ. Ο Ντέβο Στίερ πρώτο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και του δύο ομιλητέ μας. Νομίζω ότι για μας είναι άκρο σημαντικό στην Επιτροπή ανάπτυξη. μια επιτροπή που ασχολείται προφανώς με τις πολιτικές της αναπτυξιακής συνεργασίας και την ανθρωπιστική βοήθεια και σε σύγκριση με άλλες επιτροπές έχει μικρότερο λόγο σε νομοθετικές πράξεις και διαδικασίες, όμως ωστόσο κατά την άποψή μου θα πρέπει παρόλα αυτά να έχει έναν ρόλο πιο ενεργό στον έλεγχο και την άσκηση της κοινοβουλευτική διάστασης τα όσα κάνει σε σχέση με την αναπτυξιακή βοήθεια η Επιτροπή. υπ αυτήν την έννοια είναι άκρος σημαντικό, όπως είπε η Πρόεδρος αυτής της αρχής, να κατανοήσουμε και το πώς εργάζεστε, αλλά και να είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις σας για το πώς μπορούμε και εμείς να βελτιώσουμε τη δουλειά μας για την αποτελεσματική παρακολούθηση από την πλευρά του νομοθέτη του έργου της Επιτροπής. Ίσως να μην μπορούμε αμέσως, μέσα σε μία νύχτα, να υπερβούμε και να πετύχουμε την πλήρη κοινοβουλευτική παρακολούθηση της αναπτυξιακής βοήθειας από το Κοινοβούλιο, διότι δεν υπάρχει τέτοια δημοσιονομική διάσταση ακόμη, δεν είναι επισήμω ενταγμένη στον προπολογισμό. Όμω δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο νομικό για να το κάνουμε αυτό. Ήθελα λοιπόν την άποψή σα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει και το βλέπουμε και από την πλευρά του κοινοβουλευτικού ελέγχου με όλες τις πολιτικές ομάδες, ένα πολιετέ πρόγραμμα και για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αλλά σε αιτήσια βάση αυτό δεν το κάνουν όταν τα συγκεκριμένα προγράμματα καταρτίζονται. Δεν έχουμε νομικούς φραγμούς, ούτε εμπόδια που να ε, αποτρέπουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει τα αιτήσια προγράμματά της για να δούμε τα διάφορα έργα που προωθούνται. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν κατά την άποψή σας θα μπορούσε να υπάρχει ένα νέο τέτοιο επίπεδο κοινοβουλευτική παρακολούθηση και ελέγχου για να βελτιωθεί η δουλειά και αυτή τη Επιτροπή και να έχουμε τη δυνατότητα να ε, ε, έχουμε αποτελεσματικότερη παρακολούθηση αυτών των θεμάτων. Κατά δεύτερον, είπατε ότι ήσασταν το πρωί στην Επιτροπή Κόντ, ελέγχου των προπολογισμών, και θα ξέρετε ότι την ερχόμενη εβδομάδα στην μήνυ Ολομέλεια θα ψηφίσουμε τις ε, απαλλαγές Λόγου χάρη θα υποβληθεί κείμενο που θα λέει ότι το Κοινοβούλιο με μεγάλη ανησυχία σημειώνει βάσει των εκθέσεων διαχείριση το τι γίνεται με τα εκατοντάδε έργα και προγράμματα και τι πληροφορίε των αντιπροσωπιών. Τα γνωρίζετε αυτά. 45% του συνολικού ποσού των διαφόρων προγραμμάτων καθυστέρησαν, το 32% δεν έφτασαν του στόχου που είχαν τεθεί αρχικά, 29% 500 προγράμματα ή έργα έχουν καθυστερήσει ή δεν έχουν ακολουθήσει του αρχικού. Ε, επιδιωκόμενους στόχους. Θα τα γνωρίζετε όλα αυτού το είδος τα σχόλια. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν έχετε συγκεκριμένα σχόλια από αυτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας το κατέστησε σαφές ότι πιστεύουν ότι η ερμηνεία των συναδέλφων της Επιτροπής των Ελέγχων Προπολογισμών είναι λαντασμένη ως προς τους αριθμούς αλλά θέλω τη δική σας τη γνώμη. Είναι σημαντικό και για την Επιτροπή Ανάπτυξης να λάβουμε πληροφορίες από πρώτο χέρι από τους ελεγκτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο Ερίκε Γκερέρο για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και τα δύο μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου. Ιδιαίτερα χαιρετίζω εδώ τον κύριο Λένε που ήταν και συναδελφός μας για πολλά χρόνια. Ήταν πρόεδρος σημαντικής επιτροπής και πρόεδρος μάλιστα της διάσκεψης πρόεδρων επιτροπών. Είχαμε πολλές επαφές και για που ήμουν και εγώ αντιπρόεδρος των σοσιαλιστών είχαμε συχνά επαφή. Λοιπόν, θέλω να επανέλθω σε μία ιδέα που είπε και ο Νταβόρ. Δηλαδή, στην Επιτροπή μας εδώ, εμείς, πάντα διαφερόμαστε πάρα πολύ για την αποτελεσματικότητα της ε, αναπτυξιακής μας βοήθειας. Οπότε, οποιοδήποτε μέσο ελέγχου, είτε είναι επίσημο όπως είναι αυτό του ελεγκτικού συνεδρίου, είτε οτιδήποτε άλλο, συνάδει με τους στόχους της αναπτυξιακής βοήθειας που είναι ακριβώς να βοηθήσει όπως λέει και το όνομά της να βοηθήσει τους ανθρώπους που ζουν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες σε ορισμένες χώρες ώστε να μειωθούν τα προβλήματά τους που μερικές φορές αφορούν την καθημερινότητά τους και την καθημερινή τους επιβίωση. Το ελεκτικό συνέδριο λοιπόν μας βοηθάει σε αυτό το στόχο. και κάνει μέρος της δουλειάς που πρέπει να κάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι ακριβώς αυτό το monitoring. Ο έλεγχος, η εκτίμηση του πώς λειτουργούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Πάντα εισαγωγικά θέλω επίσης να πω ότι έχω περισσότερη εμπιστοσύνη στο ελεγκτικό συνέδριο και φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι εδώ επίσης από ότι σε κάποιους ευρωβουλευτές, οι οποίοι έτσι κάπως αυθόρμητα γίνονται μερικώς ελεγκτές. Μιλάω για κάποιον πρόεδρο, άντρα ή γυναίκα, επιτροπής που μερικές φορές ε, νομίζει ότι είναι μέρος του ελεγκτικού συνεδρίου. Ο Λοιπόν, έχω εμπιστοσύνη στο ελεγκτικό συνέδριο γιατί έχει τα τεχνικά στοιχεία, την ε, πληροφόρηση, ό,τι χρειάζεται για να κάνει καλά τη δουλειά του. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοηθειά σας. Τώρα για την έκθεση. Υπάρχουν πτυχές ανησυχητικές. Αναφέρονται προγράμματα, οι δείκτες, μερικές φορές δεν ορίζονται συγκεκριμένα ή λάθος. Κάτι το οποίο βέβαια επιδεινώνει τους στόχους των προγραμμάτων μας. Έχω όμως κάποιες ερωτήσεις. Έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που έγιναν τελευταία εξαιτίας της δημιουργίας αυτών ε, των ε, ταμείων ε, καταπιστημάτων. Γιατί λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από ό,τι παραδοσιακά λειτουργούν τα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας και ο έλεγχος τους εξορισμού είναι πιο δύσκολος. Εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι όντως θα είναι πιο δύσκολο να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητα και τη συμπεριφορά των ταμείων αυτών. Και θέλω να ρωτήσω και εσάς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πείτε τι γίνεται τελευταία για να βελτιωθεί η διαφάνεια. Ο κύριος Πρίνστεν, αν προφέρω σωστά το όνομά του, μας έλεγε ότι οι εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου δεν μπορεί να είναι εκθέσεις σαν να διαβάζει κανείς εφημερίδα, δηλαδή για το ευρύ κοινό, που έτσι τις διατρέχει το Σάββατο το πρωί στην πολυθρόνα του, ότι πρέπει να είναι κείμενα που να ακολουθούν κάποιους ε, κανόνες και να χρησιμοποιούν ε, και μία γλώσσα ε, που θα έλεγα τεχνική και ψυχρή. Όμως καταλαβαίνετε ότι αν η γλώσσα είναι προσιτή και την καταλαβαίνει το κοινό, τότε ενισχύεται και η διαφάνεια και όλοι οι ενδιαφερόμενοι καταλαβαίνουν καλύτερα τι λέει τελικά η κάθε έκθεσή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για να είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε τελειώσει πριν ε, το... φτάσουμε στους... στον κύριο Στυλιανίδη, παρακαλώ να είσαστε σύντομοι. Ο κύριος Γκέρεντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με τα χαράς άκουσα τον κύριο Λένε να μας λέει ότι ήταν πολύ θετικός γενικός απολογισμός. Αυτό όμως αντιφάσκει με αυτό το θόρυβο που, έχει προκαλέ, που προκαλούν συνήθω οι εκθέσει του ελεγκτικού συνεδρίου. Συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Πίνστα μόλις τώρα, ε, ότι δηλαδή η γενική αξιολόγηση είναι όπως την περιγράψατε. Και είπατε ότι δεν είστε δημοσιογράφος κύριε Πίνστα, σωστά το διευκρινίσατε. Κρίμα όμως, διότι κάποιοι δημοσιογράφοι από τις εκθέσεις σας βρίσκουν υλικό για να, κάνετε, να πετύχουν τελείως διαφορετικούς στόχους από αυτό που κάνετε εσείς με τη δεντολογία σας στο ελεγκτικό συνέδριο και ούτε θα σας είχε περάσει από το μυαλό ούτε μακράν ούτε εύκολα. Εδώ λοιπόν ήθελα να μου πείτε αν τα προγράμματα και τα έργα στα οποία αναφέρεστε τις εκθέσεις σας είναι έργα από αυστηρή έννοια ή εάν συμπεριλαμβάνεται υπό τη δημοσιονομική έννοια τα διάφορα προγράμματα. Είναι έργα ε, αυτά καθεαυτά, πολύ ωραία. Ε, είναι έργα, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι εάν ε, έχουμε τέτοια προσέγγιση για τα έργα, αυτό γίνεται γιατί δεν μπορούμε να τα εντάξουμε στον προπολογισμό. Εάν αυτό γινόταν, ε, οι δικαιούχε χώρε θα είχαν χαρακτηριστεί από την διακυβέρνησή τους για το κατά πόσον είναι ικανοί δικαιούχοι για ενίσχυση του προπολογισμό. Η παρουσίαση λοιπόν από του δημοσιογράφου των εκθέσεών σα γίνεται κατά τον εξή τρόπο. Τα έργα αυτά ε, σε έναν τόπο πιο δυσχερή, όπου υπάρχει διαφθορά, όπου η καλή διακυβέρνηση δεν είναι δεδομένη. Εάν η Επιτροπή λοιπόν σε αυτό το πολύ δύσκολο τοπίο, και εδώ πρέπει να αποτίσω φορό τιμή στην Επιτροπή που έχει τον τόλμη, να ε, επικρίνει κάποια κράτη-μέλη, διότι τι πρέπει να γίνει ε, σε αυτέ τι περιπτώσει. Τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν οι φορεί επιτόπου δεν λαμβάνουν τι σωστέ αποφάσει και καθυστερούν οι πληρωμέ. Τότε η Επιτροπή είναι πολύ υπεύθυνη στη στάση τη, λέγοντα ότι τα χρήματα δεν θα εκταμιευθούν παρά μόνο εφόσον έχουμε την εγγύηση ότι τα έργα μπορούν να λάβουν σαρκά και ωστά με τον τρόπο που θα έπρεπε. Και να πούμε ότι η διαχείριση των χρημάτων που μας ε, κατέθεσαν οι φορολογούμενοι ε, εις βάρος των οικογενειών τους, ε, η διαχείριση των χρημάτων αυτών γίνεται με τρόπο χρηστό. Εδώ λοιπόν αυτό βλέπω ότι θα θέλατε να πείτε, αν και δεν το είπατε. Είναι τελείως απαράδεκτο και σκανδαλώδες να δίνουμε έτσι επιταγές ε, εν λευκό στους λαϊκιστές όλων των προελεύσεων. Εάν λοιπόν πρόκειται για έργα δεν υπάρχει πρόβλημα. Καθυστερήσει από τον πληρωμών ε, είναι υποχρέωση για εκταμείευση αργότερα. Αυτό πρέπει να το χαιρετήσουμε και να το καταδικάζουμε. Και μετά πρέπει να κοιτάζουμε ότι βρισκόμαστε στο χείλο του γκρεμού. Διότι ε, πρέπει να είμαστε διτρέ συνετοί. Ε, η απάντηση στα προβλήματα που θα βρούμε είναι το θέμα. Εάν όλα ήταν τακτοποιημένα, θα είχαμε μόνο θετικότατε αξιολογήσει. Εάν όμω η διαχείριση ήταν όπως της Γερμανίας, της Γαλλίας ή άλλων χωρών που είναι υποδεγματικές στον τομέα αυτό, ε, το ελεγκτικό συνέδριο δεν θα είχε κανένα πρόβλημα. Θα μπορούσε να ε, αποσυρθεί κιόλα. Δεν θα είχε λόγο ύπαρξη, θα ήταν τόσο καλή διακυβέρνηση που θα περίτευε. Όμω δυστυχώ δεν ισχύει αυτό στη διακυβέρνηση αυτών των χωρών. Δεν είναι υποδεγματική. Δεν μπορούμε λοιπόν να διαφορούμε για την τύχη των χωρών αυτών. Ε, Εάν δεν θέλαμε πλέον ποτέ να εκτιθέμεθα σε αρνητικού βαθμού και αποτεμήσει, θα έπρεπε να διαφορήσουμε για την τύχη των χωρών αυτών. Θα σα τα πω πολύ ξεκάθαρα λοιπόν. Πριν ψηφίσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα, θέλω απλώ να αποκατασταθούν τα γεγονότα. Μια υπενθύμηση κάποιων αντανακλαστικών αντιδράσεων οι οποίε είναι αλληλένδετε με την χρηστή διακυβέρνηση και διαχείριση και νομίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο θα μπορούσε να πει δύο-τρία λόγια επεξηγηματικώ. Και για να μην αλλοιώνονται τα έργα και οι χειρονομίε. Διότι εγώ πραγματικά γίνομαι έξαλλο με όσα γίνονται εδώ στα πλαίσια τη αξιολόγηση και τη ερμηνεία που δίνετε στη δική σα την αξιολόγηση. Είναι πολύ ευαίσθητη διαδικασία η αξιολόγηση που κάνετε. Εάν δεν την αντιμετωπίζει κανεί με υπευθυνότητα και διοντολογία όπω ε, δει, ε, τότε δύσκολα ε, μπορεί να συνεχιστεί η πολιτική για την ανάπτυξη και βοήθεια. Κάτι που σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίστηκε στα σχόλια τη παρατηρήσης σα. Ευχαριστούμε, κυρία Χάουταλα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ χάρηκα κύριε Λένε, για την συνολικά θετική αξιολόγηση που κάνατε. Γιατί δεν εξυπηρετεί την ε, αναπτυξιακή πολιτική να γίνονται αναποτελεσματικές δαπάνες ε, ιδιαίτερα όταν η αναπτυξιακή βοήθεια χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Συγκεκριμένες ερωτήσεις τώρα. Σε ποιο βαθμό οι συστάσεις σας είναι υποχρεωτικές, δηλαδή αυτά που λέτε ε, θα οδηγήσει σε βελτίωση όταν τρέξουν τα επόμενα έργα. Θα μπορούν να αντληθούν διδάγματα για τα επόμενα έργα, δηλαδή σε ποιο βαθμό συμβαίνει αυτό. Ε, γιατί αν σκεφτώ τις εκθέσεις του ηλεκτρικού συνεδρίου για τις Γερμανίες, γιατί ε, αναφέρθηκε ότι δεν χρειάζεται εκεί, αλλά όχι, ελεγκτικό συνέδριο χρειάζεται και στη Γερμανία. Και αν δούμε τις συστάσεις εκεί και βλέποντας και ότι πολλές φορές σε συνεχόμενες εκθέσεις επισημαίνονται τα ίδια πράγματα, ε, αναρωτιέμαι αν εισακούεστε. Άλλη ερώτηση. Στην Αφρική, τα αναπτυξιακά έργα λαμβάνουν χώρα σε ε, δύσκολες συνθήκες. Σε ποιο βαθμό αυτό λαμβάνεται υπόψη στη δική σας την αξιολόγηση. Γιατί βλέπω τέσσερα σημεία, ε, ε οικονομικός ε, έλεγχος, ε, έλεγχος αποτελεσματικότητας, απόδοσης. Όλα αυτά, δηλαδή όλες τις δυσκολίες λαμβάνονται υπόψη ή ε, δεν λαμβάνεται υπόψη αυτό. Επίσης συχνά οι, τα δεδομένα και οι στατιστικές δεν επαρκούν για να γίνουν συγκριτικές μελέτες που θα καλύπτουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Αν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση στις παρεμβάσεις της ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία με βάση το αποτέλεσμα, αλλά και όταν θέλει να κάνει έλεγχο το ηλεκτρικό συνέδριο μπορεί να μην επαρκούν τα στοιχεία. Ας πούμε, ε, βελτίωση της υποδομής νηπιαγωγείων για τα παιδιά στο Μπουρούντι. Ε, αν δεν υπάρχουν δεδομένα που να καλύπτουν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πώς αξιολογούνται τα έργα στη συνέχειά τους. Θα με ενδιαφέρει αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πριν σα ξαναδώσω τον λόγο, να ακούσουμε τον κύριο Ιντολφ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρακολουθεί αυτή τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και τα δύο μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τα, για τα λόγια του. Την ίδια δουλειά κάνουμε. Θέλουμε να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα τη βοήθεια και την αποδοτικότητά τη και να προσθέσω και τον αντίκτυπο. Δεν αρχίζει με «ι» στα αγγλικά, αλλά με I, αλλά ο αντίκτυπο είναι κάτι που δεν περνάει στο, από το χέρι όποιου ε, υλοποιεί αυτή τη βοήθεια, αλλά, αλλά πολλούς άλλους ε, αλληλένδετους παράγοντες γύρω από τον τομέα της βοήθειας, μεταξύ των οποίων και η διακυβέρνηση από την ευρύτερη έννοια. Η συζήτηση από αντικατοπτρίζει αυτό που θύμισε ο κ. Πίντξτεν ότι τα πάντα έχουν να κάνουν με τη διακυβέρνηση. Η δυσκολία της εφαρμογής ε, νομοθετικών διαδικασιών, ε, με την όθηση του υπεύθυνου για την αναπτυξική βοήθεια είναι κάτι πολύ δύσκολο για να δοθούν συγκεκριμένα κίνητρα και να βελτιωθεί η διακυβέρνηση. Βέβαια, η συζήτηση αυτή πρέπει να συνεχιστεί. Και εμεί ω Επιτροπή προσφέρουμε όλη την ε, αναγκαία συνεργασία στο συνέδριο και το κοινοβούλιο για να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να εντείνουμε τις προσπάθειες βελτίωσης. Όμως το γεγονός είναι ότι πράγματι ε, λειτουργούμε σε πολύ δύσκολες ε, συνθήκες. Όχι μόνο ως προς τη διακυβέρνηση, αλλά θα φτάσουμε στο σημείο να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε με πολύ μεγάλες προσπάθειες και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Και δεν είμαι εξουσιοδοτημένος εγώ να μιλάω για όλα αυτά, γιατί ήταν μέρος της συζήτηση ευρύτερα ως προς την στρατηγική μας, ε, το στρατηγικό μας σχεδιασμό αλλά για την διευκόλυνση των χωρών ακέλογου χάρη είμαστε πολύ χαρούμενοι που η έκθεση αυτή και θέλω να προσθέσω μερικά σύντομα σχόλια. Ε, όπως ξέρετε από την ε, πλευρά μας δεν τα διαχειριζόμαστε αυτά από την ΕΤΕ τα διαχειρίζονται και είναι ένας τομέας ε, της επιχειρηματικής μας δράσης στην ανάπτυξη όπου υπάρχει κίνδυνος. Κίνδυνος να πάρουμε πρώτα τα εύκολα για να δώσουν αποτελέσματα, τα, δε, τα, τους καρπούς που είναι στα χαμηλότερα κλαδιά δηλαδή και πιο εύκολα τα πιάνουμε. Ε, τους πιάνουμε. Εδώ είπατε στο συνέδριο ότι δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να ελέγξουμε αν η ίδια χρηματοδότηση θα μπορούσε να γίνει χωρίς τις επενδύσεις. Αυτό είναι η κρίσιμη ερώτηση. θα το ε, διαπιστώσουμε μόνο με την ε, αιρεσιμότητα. Το θυμάστε, Πρόεδρε, είχαμε συζητήσει και για το blending. Ε, σε κάποιες περιπτώσεις η προσθετικότητα όπως έχει ονομαστεί είναι πολύ διαφορετική σε φτωχότερες από ό,τι σε ισχυρότερες περιοχές όπως ο ιδιωτικό τομέας που μπορεί να ενισχύσει τις παρεμβάσεις μας ενώ σε κάποιες άλλες είναι τελείως απών και έχουμε μεγαλύτερες δυσκολίες. Τι μπορούμε να κάνουμε εδώ. Ε, εδώ θα παίξει ρόλο η επικοινωνία μας προς τον ιδιωτικό τομέα όπως έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πιέσει. Επίσης με, τα, ε, χαρά ακούσαμε τα σχόλιά σας για την ειδική ενίσχυση σε πιο επικίνδυνες ε, επενδύσεις, αλλά θέλαμε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρεσορρόπηση των χωρών, διότι βλέπουμε ότι κάποιες χώρες λαμβάνουν περισσότερη προσοχή από άλλες. Ο τρόπος λοιπόν δεν είναι να είμαστε αρνητικοί στην προσέγγιση μας, απλώς να βελτιώσουμε τις ε, διαδικασίες μας, διότι η διευκόλυνση χρηματοδότησης των ΑΚΕ πρέπει να πάει βαθύτερα και να φτάσει στους φτωχότερου. Αυτό είναι ο στόχο. Είναι εύκολο στι μικρομεσαίε που ήδη τα πάνε καλά, σε μια χώρα που λειτουργεί εύρυθμα, να δώσουμε ενισχύσει. Όμω είναι πιο δύσκολο να φτάσουμε σε μια επιχείρηση, σε μια πιο δυσχερή περιοχή ή σε ένα πιο δυσχερή χώρο. Και αυτά όλα βέβαια θα επηρεάσουν και το πλαίσιο για τη νέα συμφωνία Κοτονού, όπω ξέρετε τότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά και να δούμε την ε, διευκόλυνση για τη χρηματοδότηση των ΑΚΕ. Πάντω, επαναλαμβάνω την ε, πρόσκλησή μα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι διαρκεία και καθημερινή και το λέω όχι μόνο ω ε, υπεύθυνο μάνατζερ, αλλά ω φιλόσοφο για τα θέματα αυτά. Διότι θέλουμε να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα με την δημόσια βοήθεια την οποία χειριζόμαστε. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ για, πολύ αυτέ τι διευκρινήσει τι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, όπω ακούσατε του συναδέλφου εδώ. Θέλουμε να συνεργαστούμε εντατικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δούμε όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν ξέρω ποιο θέλει να ξεκινήσει, ο κύριο ε, Πίνκτεν ή ο κύριο Λένε. Κύριε Πίνκτεν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτές μέλη τη Επιτροπής αυτής που άκουσαν πολύ προσεκτικά τα όσα είπαμε. Πολύ χαίρομαι. Και για αυτά που είπαν ο κύριος Στήρο, ο κύριος Γκερέρο, ο κύριος Γκέρενς, η κυρία Χόιμπουχ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Επιτρέψτε μου να συνοψίσω. Όσον αφορά την απαλλαγή, η συζήτηση για τα ποσά βάση της απαλλαγής στην ετήσια έκθεση δουλεύει το ελεκτικό συνέδριο, αλλά και βάσει της έκθεσης των ε, αναπτυξιακών ταμείων. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, με δύο εκθέσεις. Του EDF και την ε, δικιά σας. Και μπορεί βέβαια να έχει κάποια ένσταση η Επιτροπή, αλλά δεν συμβαίνει συνήθως. Δεύτερον, τα μέλη μας, που είναι ένας για κάθε κεφάλαιο, είναι πάντα στη διάθεση των αντίστοιχων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και πολλές φορές την πρωτοβουλία την παίρνουν ευρωβουλευτές. Εμείς περιμένουμε μέχρι να έρθουν σε επαφή οι ευρωβουλευτές με τα αντίστοιχα ε, μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Θα μπορούσε και το προσωπικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έρθει σε επαφή με το δικό μας το προσωπικό για να έχουμε τα γεγονότα και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και όπως έλεγα, δεν είναι πάντα εύκολο να διαβάσει κανείς τις εκθέσεις μας. Όντως, εμείς πρέπει να ανταποκριθούμε στις προδιαγραφές. Έχουμε μια διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι ο κανονικός έλεγχος. Ο ελεγχόμενος έχει το δικαίωμα να απαντήσει και να συμφωνήσουμε τα ποσά. Αν έρθει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας δώσει καλύτερα στοιχεία από αυτά που έχουμε εμείς, εμείς τους λέμε μάλιστα ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Τίποτα παραπέρα. Τώρα βέβαια εννοείται ότι δεν αντικαθιστούμε εμείς τους ευρωβουλευτές. Αν στην Ολομέλεια εσείς αποφασίσετε για, το δικό σας, για τη δικιά σας απαλλαγή, για το έγγραφο απαλλαγής, εμείς σας δίνουμε ό,τι πληροφορίες έχουμε και εσείς ευρωβουλευτές αυτόνομα αποφασίζετε. Συνήθως λαμβάνετε υπόψη τις παρατηρήσεις μας και τα στοιχεία που δίνουμε. Αυτά για την απαλλαγή αλλά και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως σε κάθε κοινοβούλιο, η συζήτηση για την απαλλαγή είναι μια δύσκολη συζήτηση και λεπτή, από την οποία απορρέουν διάφορες διστάμενες απόψεις. Πάντα συμβαίνει αυτό και πάντα θα συμβαίνει και στο μέλλον. Ένα είναι αυτό. Τώρα για τις νέες ε, δημοσιονομικές τεχνικές. Σήμερα το πρωί κάποιος με ρώτησε, όταν αναφερόμουν στην αναθεώρηση ε, κινδύνου, στα πλαίσια των Panama Papers, το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι κάποια στιγμή αυτού του είδους οι πληροφορίες που έχουμε για τις τράπεζες, τα Panama Papers, κάπου να έχουμε νέα μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται αλλά που δεν χρησιμοποιούνται όπως θα έπρεπε. Και με ρώτησαν, έχετε καμιά τέτοια ένδειξη. Όχι, δεν έχω. Η Επιτροπή σίγουρα είναι πολύ προσεκτική, αλλά αν υποθέσουμε ότι επιλέξει κάποιο μηχανισμό θα πρέπει να το σκέφτεται δύο φορές παραπάνω από ότι οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα. Και είμαι σίγουρη ότι το κάνουν. Γιατί όσο πιο περίπλοκοι είναι οι μηχανισμοί, τα μέσα που χρησιμοποιούνται, τόσο βέβαια μεγαλύτερη είναι η μόχλευση, αλλά τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα διευθυντικά ταμεία, όλοι τέλο πάντων, πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ πώς δαπανούν τα κονδύλια του προπολογισμού. Και έτσι έρχομαι και στο στοιχείο του κινδύνου. Πιστεύω ότι αν δαπανά κανείς χρήματα, και πόσο μάλλον στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας, δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος. Πάντοτε θα ελοχεύει κάποιος κίνδυνος. Και πολύ συχνά στις ειδικέ μας εκθέσεις αναφέρουμε τους κινδύνους αυτούς και λέμε ότι εξαιτία της πολιτικής αστάθειας, για παράδειγμα, ή εξαιτία διαφθοράς, υπάρχει κίνδυνος. Δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος δηλαδή. τα προγράμματα ε, στήριξη του προπολογισμού, συνεργασία με τον ΟΗΕ, με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό το οποίο πάντα τονίζουμε είναι ότι πριν χρησιμοποιηθεί κάποιος μηχανισμός, θα πρέπει να προηγείται ανάλυση. Γίνεται αυτό πάντα? Όχι, δεν γίνεται και μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα με τον ε, αγαπητό συνάδελφο Κλάους Λένε συζητήσαμε για ένα έγγραφο της Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την βοήθεια στη Μολδαβία. Μπορείτε να το διαβάσετε αργότερα το έγγραφο άμα θέλετε, αλλά τι λέει, λέει ότι μερικές φορές οι, οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται, αλλά την ίδια στιγμή καλύπτονται. Ωραία. Το λέμε στο έγγραφο. Και από εκεί και πέρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ό,τι νομίζει. Πάντως σε πολλές περιπτώσεις οι προϋποθέσεις είχαν ήδη καλυφθεί. Παρόλα αυτά εμείς το αναφέραμε στην έκθεσή μας. Αυτό θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι χρηστή η οικονομική διαχείριση, για να το πω έτσι πια. Μερικές φορές δηλαδή είμαστε αντιμέτωποι με πράγματα που γίνονται, το συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι δεν είναι όλα τέλεια. Και τελειώνω με το εξής με τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε στη διατύπωση. Όλα αυτά που κάνουν τα μέλη του λεκτικού συνεδρίου έχουν να κάνουν με τον τρόπο με τον οποίο κρίνονται τα πράγματα. Τα μέλη του λεκτικού συνεδρίου πρέπει να είναι δίκαια Άρα πρέπει να έχουν τα προσόντα για να το κάνουν. Την ποιότητα δηλαδή. Γιατί αυτό είναι που μένει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στους τίτλους των εφημερίδων. Άρα πρέπει να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Όπως ακριβώς πρέπει και οφείλουμε. Ο κύριος Λένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να συμπτύξω τις απαντήσεις όταν ε, μιλάμε για αναπτυξιακή βοήθεια, εγώ ασχολούμαι στο τρίτο τμήμα εδώ και δύο χρόνια, δύο-τρία χρόνια, υπάρχουν τρεις μηχανισμοί. Το ένα είναι η επιδότηση των έργων, έχω ένα έργο δηλαδή και δίνω κονδύλια ευρωπαϊκά για να πραγματοποιηθεί. Ο άλλος τρόπος είναι η δημοσιονομική υποστήριξη άμεσα από τον προϋπολογισμό σε ένα κράτος, ούτω ώστε να μπορεί να ακολουθήσει μια πολιτική και να την εφαρμόσει. Και το τρίτο που μας απασχολεί εν προκειμένου είναι η διάθεση κεφαλαίων, είτε μέσω ε, δανείων ή ε, συμμετοχών επενδυτικών για να γίνουν κάποια έργα. Νομίζω ότι και τα, οι, τρεις, τα τρία, οι τρεις αυτοί μηχανισμοί έχουν λόγο ύπαρξης οι διαφορετικές μεθοδολογίες μπορεί να εξυπηρετούν κάποια στιγμή σε ορισμένε περιπτώσεις, αλλά όχι σε όλες. Μπορεί πολλές φορές να συνεπάρχουν οι διαφορετικές μεθοδολογίες, αλλά ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την χορήγηση δανείων πρέπει να προηγηθεί πολύ σημαντικός έλεγχος εκ των, προ... εκ προτέρων, ούτως ώστε να ελεγχθεί η απόδοση, η αντίκτυπος, αποτελεσματικότητα κτλ. Ε, εδώ τα είχαμε πάει καλά στην ε, έκθεση. Πολλές φορές πρέπει να συντονίζουμε τις ε, ενέργειές μας και με άλλους, όπως με την Κομισιόν, για να εξετάσουμε το νόημα που έχουν τα οι ε, είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σε περιοχές ε, φτωχές, κυρίως της Αφρική, γιατί εκεί γίνονται περισσότερα έργα, να γίνεται αυτός ο έλεγχος. Ε, με τις επιδοτήσεις, πολύ σημαντική είναι η παρακολούθηση. Δηλαδή, όταν ε, ε χορηγούνται επιδοτήσεις, ε, ιδιαίτερα όταν γίνεται η πληρωμή με δόσεις, θα πρέπει να παρακολουθούμε αν τα έργα εξελίσσονται όπως πρέπει και στη δημοσιονομική στήριξη και εκεί η παρακολούθηση, το monitoring είναι πολύ σημαντικό γιατί θα πρέπει να δούμε τι ε, κάνουν οι κυβερνήσεις, η κάθε κυβέρνηση που θα ε, πάρει τα κονδύλια. Ε, μπορεί ε, όλες οι μέθοδοι να οδηγήσουν σε επιτυχία. Υπάρχει ένας παράγων που δεν επηρεάζεται εύκολα και έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες κάθε φορά. Είναι ο ανθρώπινος παράγων. Μπορεί να κάνετε τέλειο σχεδιασμό. Αν επί τόπου δεν είναι σωστό το ανθρώπινο δυναμικό που θα ε, υλοποιήσει το πρόγραμμα, ε, όχι μόνο εξειδίκευση, αλλά επικοινωνιακές δεξιότητες, ανθρώπινες ικανότητες. Αν δεν υπάρχουν αυτές, δεν θα ε, υπάρχει επιτυχία. Ο ανθρώπινος παράγων είναι καθοριστικός. Αλλά ε, αυτόν ε, περιορισμένα τον επηρεάζουμε. Τώρα, για τα δεδομένα. Πάντα πρέπει να είναι ασφαλή τα δεδομένα. Πώς θα κάνουμε έλεγχο αν δεν έχουμε ασφαλή δεδομένα. Όμως υπάρχει πληθώρα πηγών, το ξέρετε πολύ καλά, που μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Καμιά φορά η αξιοπιστία είναι λίγο περιορισμένη, αλλά άμα συγκρίνουμε τη μία πηγή με τις άλλες, Μπορούμε έτσι να έχουμε ασφαλή στοιχεία και να τα χρησιμοποιούμε. Τώρα, το ε, θέμα των media, νομίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο τα προηγούμενα χρόνια έκανε κινήσεις τέτοιες ώστε να βελτιώσει την εικόνα του στα media. Και αυτό το έκανε με τρόπο επαγγελματικό. Δηλαδή, εμείς κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αποφεύγουμε, να εκπέμπουμε λάθος μηνύματα. Από την άλλη, καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που συνειδητά θέλουν να διαδώσουν λάθος μηνύματα και μετά να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα για δικούς τους σκοπούς. Ε, παραπλάνηση για ίδιους σκοπούς. Εμείς, όπως είπε και ο κύριος Πίνξτεν, ε, έχουμε πολύ ξεκάθαρη μεθοδολογία όταν καταρτίζουμε τις εκθέσεις μας. Είμαστε υποχρεωμένοι γι' αυτό. Θα μπορούσαμε να είμαστε πιο φιλικοί προς τον αναγνώστη. Από την άλλη όμως είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που πρέπει να παρουσιάσουμε και αυτό οδηγεί σε ένα φορμαλισμό που ως ένα βαθμό είναι αναπόφευκτος. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές μας για την τόσο καλή επισκόπηση που μας έδωσαν, το τόσο υλικό για σκέψη. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε καλύτερα και τη δουλειά σας και πώς μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε μαζί σας. Νομίζω ειλικρινώς ότι ε, με τη γραπτή διαδικασία έχουμε διαρκώ επαφέ με το ελεγκτικό συνέδριο. Οι δικοί μα εισηγητέ μιλούν με του δικού σα ειδικού εισηγητέ. Αλλά πραγματικά η συζήτηση αυτή είναι χρήσιμη για να καταλάβουμε καλύτερα τι κάνετε και, και εσεί να ετοιμάζετε καλύτερε εκθέσει και εμεί να κατανοούμε καλύτερα το τι κάνετε. Σα ευχαριστούμε.

Sorry, colleagues, we're just look waiting. Συνάδελφοι, περιμένουμε τον Επίτροπο. Σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσουμε να δούμε τι του έχει συμβεί.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 colleagues, can people now take... Συνάδελφοι, παρακαλώ καθίστε. Πριν ε, περάσουμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 17, θα ήθελα επισήμω να καλωσορίσω αντιπροσωπεία ε, υπαλλήλων από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο που κάθονται εδώ στην ε, τρίτη σειρά από το τέλο. Καλωσορίζω ολόκληρη την αντιπροσωπεία τον κύριο Γιουσούφα Κτού ε, στην τελευταία ημέρα μια τρίμερη επισκεψή του στο Κοινοβούλιο. Ε, δουλειά μας είναι να παρακολουθήσουμε το Παναφρανικό Κοινοβούλιο στην προσπάθειά του να περάσει από ένα συμβουλευτικό σώμα σε ένα νομοθετικό. Ε, είναι μια διαδικασία δύσκολη, βαθμία. Εργάστηκα εδώ και την δεκαετία του 80 και εμεί ήμασταν ε, συμβουλευτικών αρμοδιότητων ηθικά. Μετά αναλάβαμε νομοθετικέ αρμοδιότητε. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει αλλάξει πολύ το κοινοβούλιο το δικό μα και με τα χαράζει να ανταλλάξουμε εμπειρίε μαζί σα. Όλα αυτά τα διοργάνωσε η ομάδα για τον συντονισμό και την προώθηση της δημοκρατίας που συντονίζουμε με τον κύριο Μπροκ. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας λοιπόν. Σας ευχαριστούμε για την επισκεψή σας και αν έχετε απορίες μετά την τέλος της συνεδρίασης μπορείτε να έρθετε να μας δείτε. Ξέρετε που είμαστε πλέον. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα στο σημείο 17, στον διευθυνμένο διάλογο σχετικά με το πρόγραμμα εργασία τη Επιτροπή και καλωσορίζουμε τον Επίτροπο Στυλιανίδη, Επισήμω οι, η επιτροπή μα επισκέπτονται τουλάχιστον άπαξ ετησίω, αλλά εσεί έρχεστε συστηματικότατα στην επιτροπή μα. Είμαστε πραγματικά εξοικειωμένοι με τη δουλειά σα. Ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνετε, διότι διαρκώ τα βλέπω στο BBC, στις ειδήσει. Την περασμένη εβδομάδα σα είδα στην Αιθιοπία και για την, να μιλάτε στην Αντίσα Μπέμπα για την ξηρασία που επικρατεί στη χώρα. Στα πλαίσια του διαφθορμένου διαλόγου, λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα εργασιών τη Επιτροπή για φέτο, αλλά και το τι προγραμματίζεται για του χρόνου, τι θα πρέπει να γίνει του χρόνου. Τα πορίσματα του διαλόγου τα γνωστοποιούμε στην διάσκεψη των, επιτροπών, των Προέδρων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και τη διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου για να ληφθούν και σχετικέ αποφάσει ειδικέ μα για το πρόγραμμα εργασία τη Επιτροπή το 2017. Δεν θα σα καθυστερήσω παραπάνω. Το 2016 και σε άσχημα. Τι να σα πω τώρα, θα έκανα του χρόνου. Αν και καλύτερα πάντοτε κανείς να προγραμματίζει γέρος. Πάντως τις ερχόμενες εβδομάδες έχουμε μια σημαντική εκδήλωση την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη τον Μάιο και ξέρουμε ότι θα οδηγήσει σε, κάποια, σε κάποιο επαναπροσδιορισμό της ανθρωπιστικής βοήθειας. Με τα χαράς λοιπόν να σας ακούσουμε και να μας πείτε τι έγινε στις πιο πρόσφατες επισκέψεις σας γιατί από εκδρομές μαθαίνει κανείς πολλά τελικά από αυτές τις επιτόπιες ε, διαπιστώσεις του πώς έχουν τα πράγματα. Ο λόγος εσά λοιπόν. Σε ευχαριστώ Λίντα, ευχαριστώ. Ε, ορίζω τους φίλους μας από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και εγώ. Και θα ήθελα να πω ότι η εμπειρία μας στην Αιθιοπία τις περασμένες εβδομάδες, ιδίως σε μια περιοχή που έχει πληγεί από το Ελληνίνιο, ήταν πραγματικά πολύ επώδυνη, πολύ δυσάρεστη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχουν προβλέψει ένα σημαντικότατο ποσό για να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης εκεί. Συνάδελφοι, είναι πολύ ευχαριστώ να σας ξαναβλέπω λίγες εβδομάδες μόλις μετά την τελευταία μας συνάντηση. Έχουν συμβεί πραγματικά σημαντικά πράγματα τις τελευταίες αυτές εβδομάδες. Και είναι μεγάλη μου χαρά να μπορώ να τα συζητήσω μαζί σας. Πάντοτε σε ένα κλίμα θετικό και βέβαια σχολιάζοντας ταυτόχρονα και την εφαρμογή των επιχειρησιακών μας προτεραιοτήτων καθώς και τις νέες και να εξελίξει πολιτικές μας πρωτοβουλίες. Θα ήθελα επίσης να σχολιάσω την ε, επερχόμενη ε, Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Τον περασμένο μήνα εκπροσώπησα και παρουσίασα το νέο εργαλείο για έκτακτη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός του, της επικράτειας της Ένωσης. Είναι μεγάλη μου χαρά σήμερα να μπορώ να ανακοινώσω έναν μόλις μήνα μετά την εξαγγελία ότι τα οι πρώτες οκτώ συμβάσεις έχουν ήδη υπογραφεί. Χθε μετέβουν προσωπικό στην Αθήνα για να προβώ σε αυτή την εξαγγελία μαζί με τις ε, ελληνικές αρχές και τους ε, υπευθύνους για ανθρωπιστικές υποθέσεις. Αυτή η διαδικασία, η επιταχυμένη, ε, αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση νοιάζεται και ότι μπορεί να αναλάβει δράση γοργά. Μας χρειάστηκε μόλις ένας μήνας από τη στιγμή που υποβλήθηκε η πρόταση έως την πραγματική παροχή βοήθειας και στήριξης είναι μοναδικό ε, γεγονός ε, για τη δράση των θεσμικών οργάνων. Χάρη και στη δική σας βοήθεια και την επικοδομητική σας προσέγγιση όλα αυτά. Η συντριπτική πλειοψηφία που στήριξε τον διορθωτικό προπολογισμό την περασμένη εβδομάδα για τα πρώτα 100 εκατομμύρια ευρώ ήταν πραγματικά μια ισχυρότατη πολιτική στήριξη. Προφανώς πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η στήριξη αυτή θα παρασχεθεί βάσει με τα υψηλά μας πρότυπα. Γι' αυτό πρέπει να εργαστούμε με, έμπειρους, με έμπειρες και οικονομικώς βιώσιμες ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι οποίες έχουν ήδη συμφωνίες συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι υπηρεσίες μου, Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ και εγώ θα παρακολουθούμε στενά αυτές τις προσπάθειες για να διασφαλίσουμε την ποιότητά τους. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη αποσταλεί υπαλληλικό προσωπικό στην Αθήνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε ότι η κρίση των προσφύγων είναι συνέπεια της ε, σοβαρότατης ανθρωπιστικής κρίσης, των κρίσεων που απαντώνται να τον κόσμο. Είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο που απαιτεί παγκόσμια και συνολική απάντηση και αντιμετώπιση. Το Σάββατο βρισκόμουν στην Τεχεράνη μαζί με μια αντιπροσωπεία Ευρωπαίων Επιτρόπων, τον οποίον ηγείτο η ύπατη εκπρόσωπος, η κυρία Φεντερίκα Μογκερίνη. Εκεί εξήγηλα αυξημένη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 3 εκατομμύρια Αφγανούς πρόσφυγες στο Ιράν. Είχαμε επικοδομητικές συνομιλίες και προτίθεμε να έχω κι άλλη επίσκεψη εκεί, να οργανώσω κι άλλη επίσκεψη εκεί τον Ιούλιο. Βάσει τη είπα τη αρμοστία του ΙΕ για του πρόσφυγε, αυτή τη στιγμή πολλοί Αφγανοί που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη περάσει κάποιο διάστημα στο Ιράν στο παρελθόν. Αυτό το επιπλέον παράδειγμα δείχνει ότι η κρίση των προσφύγων έχει διεθνή και διακρατικό χαρακτήρα. Ταυτόχρονα η συνολική, η σφαιρική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό απαιτείται πλέον. Να ε, σχολιάσω τώρα τις μεγαλύτερες ε, κρίσεις ανθρωπιστικού χαρακτήρα και τις πρόσφατες εξελίξεις για να δείτε τι κάνουμε στην, στο επικλησιακό επίπεδο. Στη Συρία, η εκχειρία που συμφωνήθηκε το Φεβρουάριο είναι ευάλωτη και δέχεται διαρκώς μεγαλύτερες πιέσεις. Το γνωρίζετε. Ξέρετε τι γίνεται γύρω από το Χαλέπι. Μερικά στοιχεία μόνο. Πάνω από 200.000 άνθρωποι έχουν ε, εκτοπιστεί ήδη από τον Φεβρουάριο και μόνον. Ταυτόχρονα η πρόσβαση σε πολυερκούμενες περιοχές παραμένει δυσχερής. Από την ε, στιγμή που ξέσπασε αυτή η κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικώς έχει ε, εκταμιεύσει και δεσμεύσει 5,7 δις ευρώ για ανθρωπιστική αναπτυξιακή βοήθεια και βοήθεια σταθεροποίησης. Γνωρίζετε ότι στη Σύνοδο του Λονδίνου για την κρίση της Συρίας στις 4 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι ε, ε, δεσμεύτηκε περισσότερο από όλους. 2,4 δις για το διάστημα 2016-2017. Από αυτά τα 2,4 δις 445 εκατομμύρια ευρώ είναι πρόσθετη ανθρωπιστική στήριξη προ τη Συρία, την Τουρκία, το Λίβανο και την Ιορδανία μόνο για το 2016, την τρέχουσα χρονιά. Από τη δική μας την πλευρά εκταβιεύουμε ποσά για την ανθρωπιστική διάσταση τη διευκόλυνση προσφύγων στην Τουρκία. Τα πρώτα 90 εκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη δεσμευτεί. Άλλα 75 εκατομμύρια θα ε, εκταμιευθούν έως τα μέσα Ιουλίου. Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πλήρως αφοσιωμένη στο στόχο να βρεθεί πολιτική λύση στο πρόβλημα. Στηρίζουμε 100% τις προσπάθειες του ειδικού επιτετραμένου του ΙΕ Στέφανο Ντεμιστούρα για το θέμα αυτό και επίσης συμμετέχουμε ενεργά στις εργασίες της Διεθνούς Ομάδας Υποστήριξης για τη Συρία. Κάθε ομάδα κρούσης ανθρωπιστικού χαρακτήρα διευκολύνει τόσο την πρόσβαση όσο και την παροχή βοήθειας που τόσο πολύ χρειάζεται η Συρία. 450.000 άνθρωποι ε, έλαβαν βοήθεια σε πολιορκούμενες περιοχές φέτος μόνον. Μεγάλο επίτευγμα σε αυτό στις τόσο δύσκολες και αντίξωες συνθήκες. Αυτό, ωστόσο, το, αυτός ο αριθμός ε, εκπροσωπεί μόνο το 10% όλων των σύρων που χρήζουν βοήθειας. Πρέπει να εντείνουμε τις προσπαθίες μας, όχι μόνο από την ε, χρηματική σκοπιά, αλλά επειδή πρέπει να προάγουμε και τα συμφέροντά τους. Στο Ιράκ τώρα. Η δέσμευσή μας ως προς τη Συρία πρέπει να συμβαδίσει με παρόμοιες δεσμεύσεις για το Ιράκ. Οι ανθρωπιστικές ανάγκες εκεί είναι τεράστιες. 10 εκατομμύρια άνθρωποι χρήζουν βοήθεια. 3,4 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί εσωτερικώς. Ο αντίκτυπος των εξελίξεων στο Ιράκ στην ευρύτερη περιοχή και πέραν αυτών των ε, γεωγραφικών ορίων είναι καθοριστική σημασία. Θυμηθείτε, το Ιράκ είναι η τρίτη χώρα αφήξεων μεταναστών προς την Ευρώπη. Τρίτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και εδώ πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανθρωπιστική απόκριση που θα βρούμε στο πρόβλημα αυτό. Μόνο πέρσι ε, μπορέσαμε να δώσουμε πάνω από 500 εκατομμύρια, 105 μάλλον εκατομμύρια ευρώ και καλούμε για την προστασία του άμαχου πληθυσμού των πολιτών καθώς και για τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και για την ανθρωπιστική πρόσβαση. Πάνω από 84 εκατομμύρια ε, ευρώ ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιήθηκαν φέτος ε, για το Ιράκ, μεταξύ των οποίων 5 εκατομμύρια για την ε, εκπαίδευση για επίγουσες, καταπήγουσες ανάγκες. Η Εμένη. Η Εμένη σήμερα είναι σε πολύ μεγάλη κρίση, ανθρωπιστική κυρίως. Και μάλιστα σε ρυθμούς απόλυτους πάνω από 21 εκατομμύρια ε, άνθρωποι χρειάζονται βοήθεια. 21 εκατομμύρια. Πάνω από 10% του πληθυσμού αυτή τη στιγμή έχουν εκτοπιστεί εσωτερικώ. Και αντιμετωπίζουμε, όπως ξέρετε, τεράστιε δυσκολίες για να παράσχουμε ανθρωπιστική βοήθεια στην Ιεμένη. Η εκεχηρία είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Αλλά πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε στις διάφορες πλευρές τις πλευρές της ε, διένεξης, ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, δηλαδή να επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση. Και βεβαίως για να υπάρξει η εφαρμογή των διατάξεων σε σχέση με τη διάσωση ανθρώπινων ζώων και να σέβονται και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Ουκρανία. Με την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Ανατολική Ουκρανία, για πρώτη φορά Ε, επισκέφθηκα μια περιοχή όπου πραγματικά ανθρώπινο πόνο δεν βρίσκεται πλέον στον ε, μικροσκόπιο των διεθνών ε, μέσων ενημέρωσης. Να σα τα πω ξεκάθαρα. Η κρίση στην Ουκρανία είναι κάτι που δεν μπορούμε να παραβλέπουμε. Πάνω από 3 εκατομμύρια χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Επανεπιβεβαίωσα την πλήρη αλληλεγγύη που θα επιδείξει η Ευρωπαϊκή Ένωση προ το λαό τη Ουκρανία και ανακοίνωσα ε, επιπλέον στήριξη πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ για φέτο μόνον, λέγοντα και πάλι ότι αυτό συμπεριλαμβάνει πάνω από 2 εκατομμύρια για την ε, εκπαίδευση σε έκτακτε ανάγκε. Επικεντρώνομαι σε αυτά διότι είδα ότι είναι ένα σημαντικότατο εργαλείο αυτό για να βελτιωθεί η κατάσταση των παιδιών, η συνθήκη ζωή των παιδιών. Δυστυχώ, ένα χρόνο μετά την υπογραφή τη συμφωνιών του Μίνσκ, η ειρήνη και η σταθερότητα δεν έχουν αποκατασταθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να καλεί όλε τι πλευρέ να σέβονται αυστηρό την εκεχηρία επανέλαβα τις εκκλήσεις μας προς όλες τις πλευρές να επιτρέψουν την ε, δίχως ε, προσκόμματα πρόσβαση στους ε, φορείς ανθρωπιστικής βοήθειας. Η άρνηση πρόσβασης και η αναστολή ανθρωπιστικών δράσεων από τις αποκαλούμενες αρχές στις περιοχές που δεν ελέγχει η κυβέρνηση είναι απαράδεκτη. Νότιο Σουδάν, Πραγματικά εδώ έχουμε τον ορισμό της αποτυχίας ε, των φορέων της διεθνούς κοινότητας να πετύχουν σταθεροποίηση της περιοχής. Είναι ντροπή μας. Στο Νότιο Σουδάν ένας θανατηφόρος πόλεμος συνεχίζει να οδηγεί στην απώλεια ανθρώπινων ζώων. Μιλάμε για φόνους αδιακρίτως, για βιασμούς, λοιμό και εκτοπισμούς. Το ξέρετε καλύτερα από εμά. Ξέρετε ποια είναι η κατάσταση εκεί, συνάδελφοι. Οι ηθήνοντες αυτής της χώρας πρέπει να σεβαστούν επιτέλους τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και να προστατεύουν τους ε, πολίτες, τον άμαχο πληθυσμό. Πρέπει να λογοδοτήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ό,τι μπορεί για να διευκολύνει την θέσπιση και την ε, εγκαθίδρυση μιας μεταβατικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας και μόλις αυτό επιτευχθεί θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε έναν ειλικρινή διάλογο των επιχειρησιακών για να χτίσουμε το μέλλον της χώρας. Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτό το σκέλος της παρουσίασής μου με μία αναφορά στην κρίση του ιού έμπολα. Ένα από τα βασικά διδάγματα που αποκομίσαμε ήταν η επίγουσα ανάγκη να βελτιώσουμε τις διεθνείς μας δυνατότητες, τις δυνατότητες μας μάλλον διεθνώς, για να παράσχουμε ιατρική βοήθεια. Ε, πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότητες της Ευρώπης να αντιδράσει σε εκτακτά περιστατικά υγείας. Υπήρξαμε μάρτυρες νέων κρουσμάτων του έμπολα και αυτή η νέα δυνατότητα πρέπει να ε, βρεθεί ε, άμεσα διότι παραμένει απαραίτητη. Βεβαίω ευτυχώ ελέγξαμε την κατάσταση. Αλλά δεν μπορούμε να πάψουμε να επαγρυπνούμε. Με την ε, Είμαι υπερήφανος διότι ήδη ε, ιδρύσαμε το Ευρωπαϊκό Ιατρικό Σώμα τον περασμένο Φεβρουάριο και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε επιτέλους ότι μπορεί να παράσχει χειροπιαστές λύσεις σε προβλήματα διεθνούς κλίμακας. Επιτρέψτε μου τώρα να στραφώ στις νέες και διαρκείας ε, πολιτικές πρωτοβουλίες, πολιτικές Να ξεκινήσω με τις πρώτες μας προτεραιότητες που είναι και δικές μου. Όπως σας είπα είναι δική μου αιμονή η κατάρτιση και η εκπαίδευση για τις ε, έκτακτες συνθήκες. Πέρυσι δεσμεύτηκα να αυξήσω την ανθρωπιστική βοήθεια από 1 σε 4% για την εκπαίδευση σε έκτακτες ανάγκες. Περίπου 40 εκατομμύρια παιδιά αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνουν ε, σχολείο σε περιοχές που έχουν πληγεί από κρίση περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν να μην τελειώσουν τις σπουδές τους, τη θήτησή τους. Δεν μπορούμε απλώς να παραμένουμε αδιάφοροι. Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μορφωθεί. Το να επενδύσουμε στην παιδεία τους, και το πιστεύω ακράδαντα αυτό, είναι επένδυση στο μέλλον τους. Πετύχαμε το στόχο μας, μαζί Πριν από λίγες ημέρες εξήγηλα την ε, δέσμευσή μας ε, την πίστοση του προπολογισμού για φέτος και μόνον. Από 11 εκατομμύρια πέρσι προβλέπουμε φέτος 52 εκατομμύρια ευρώ για το 2016. Αυτό ξεπερνά ακόμη και τον στόχο του 4% που είχαμε θέσει. Το ίμιση αυτού του ποσού προέρχεται από το διευθυντικό του προπολογισμού που η επιτοπή σα επιτυχώς πρότεινε και το συνολικό ποσό είναι σε κάθε περίπτωση ε, άκρος συμβολικό, διότι αποδεικνύει τις κοινέ μας προσπάθειες, την επιτυχία μας, το πώς Επιτροπή και Κοινοβούλιο είμαστε χέρι-χέρι στον αγώνα αυτό και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την δική σας πυγμή και αποφασιστικότητα στην κοινή μας αυτή πρωτοβουλία. Με αυτό το πακέτο θα πετύχουμε να καλύψουμε τις ανάγκες πάνω από 2 εκατομμυρίων 300 χιλιάδων παιδιών σε 42 χώρες. Τα προγράμματα που θα επιλεγούν θα καλύψουν τις ανάγκες παιδιών που έχουν πληγεί από διενέξεις και πόλεμο και την πρόσβασή τους σε ποιοτική εκπαίδευση. Ιδίω για την κρίση στη Συρία. Οι δράσεις μας θα συμπληρώσουν αυτές που χρηματοδοτούνται από άλλες υπηρεσίες τη επιτροπή. Θα επικεντρωθούν κυρίως στις δραστηριότητες άτυπη εκπαίδευση. όπως την εκπαίδευση για τον κίνδυνο από τις ε, νάρκες, τις ε, δεξιότητες ζωής και την επαγγελματική κατάρτιση. Έχω πολλές τέτοιες εμπειρίες σχετικά. Είδαμε να γίνεται ήδη πολύ καλή δουλειά από τους συνεργάτες μας και είδα τα παιδιά να είναι πραγματικά χαρούμενα με αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, με τη στήριξη που τους δίνεται για την εκπαίδευσή τους. Φέτος θα επικεντρωθούμε επίσης στην άτυπη εκπαίδευση των ε, Αφγανών μεταναστών στο Ιράν. Σας ε, παρουσίασα το πρόγραμμά μας, το προσεχές μας πρόγραμμα με τους εταίρους μας και το συζήτησα και πριν από τέσσερις ημέρες στην Τεχεράνη. Επίσης θα παράσχουμε στήριξη στα παιδιά της λίμνης Τσάντ, της περιοχής αυτής που ε, προσπαθούν να ξεφύγουν από τον Μπόκο Χαράμ, την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και τις υπηρεσίες προστασίας των παιδών. Επίση, θα επικεντρωθούμε στην εκπαίδευση των μεταναστών στην Τουρκία. Όχι μόνο στην Τουρκία, μάλλον, αλλά και στην Ελλάδα. Θα προβλεφθούν για το σκοπό αυτό επιπλέον 52 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτηθούν τα σχετικά προγράμματα. Δεύτερη προτεραιότητά μα είναι να αντιμετωπίσουμε τον εκτοπισμό μακρά διαρκεία. Μαζί με του ε, αγαπητού μου συναδέλφου, την Φεντερίκα Μογκερίνη και του επιτρόπου Μίμητσα και Χάν, ε, περατώνουμε μια ανακοίνωση για, την, ε, για τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό και την ανάπτυξη. Αυτή θα ε, ε, σας υποβληθεί στο τέλος του μήνα. θα έχουμε συγκεκριμένους πολιτικούς προσανατολισμούς και καθοδήγηση για το πώς οι φορείς πολιτικής, ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας μπορούν να συνεργαστούν με τοπικές κοινότητες και κυβερνήσεις. στο ξέσπασμα μιας κρίσης εκτοπισμού με έναν τρόπο στρατηγικό και σφαιρικό. Θέλουμε να πάψει η εξάρτηση για τη βοήθεια και να αναπτυχθεί η ανεξαρτησία των μεταναστών και των ανάλογων φορέων. Θέλουμε να αποκατασταθεί η αξιοπρέπειά τους και να τους δώσουμε ελπίδα. Η προτεραιότητα αυτή είναι ο τρόπος που έχουμε βρει να συνδέσουμε την ανθρωπιστική και την αναπτυξιακή συνιστόσα επιτόπου. Η τρίτη μας προτεραιότητα είναι η ανθεκτικότητα. Το να αναπτύξουμε αντοχή και ανθεκτικότητα σημαίνει ότι θα επικεντρωθούμε στην πρόληψη και την ετοιμότητα. Η αναχέτηση και η μείωση των κινδύνων είναι ζωτική σημασίας. Η Επιτροπή θα εγκρίνει τι προσεχεί εβδομάδε το πρόγραμμα δράση για την εφαρμογή των προτεραιοτήτων που αναλήφθηκαν στο ΣΕΝΤΑΙ για την μείωση των κινδύνων από καταστροφέ είναι μια καλή ευκαιρία για να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα. Το πρόγραμμα αυτών δράσης θα θέσει τα θεμέλια για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης για την ενημέρωση περί κινδύνων και θα μεταφράσει τις προτεραιότητες αυτές στο πλαίσιο του ΣΕΝΤΑΕ και θα τις απλώσει σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως σας είπα, επιστρέφω από την Αιθιοπία. Επέστρεψα πριν από λίγες ημέρες και μπορώ να σας μιλήσω για τι σοβαρότατε βλάβες που έχω προκαλέσει το Ελνίνιο. Η επισητιστική ε, ανασφάλεια αυτή τη στιγμή επηρεάζει 20 εκατομμύρια ανθρώπους εκεί. 20 εκατομμύρια. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το πρόσθετο πακέτο 122,5 ε, εκατομμυρίων ευρώ για ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια. Με τον Εύεν Μίμητσα ψάχνουμε τρόπους για να συνεργαστούμε και να καλύψουμε ανάγκες που μπορεί να απειλούν την ίδια την επιβίωση των ανθρώπων εκεί, αντιμετωπίζοντας βεβαίως ταυτόχρονα και τα γενεσιουργά αίτια. Δυστυχώς τέτοια φαινόμενα απλώς θα πολλαπλασιάζονται στο μέλλον. Έχουμε συλλογική ευθύνη, συνάδελφοι, να δράσουμε. Πρέπει να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και να είναι έτοιμοι οι ίδιοι με δική τους αντοχή να αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά και αυτή είναι και η στόχη που αναλάβαμε στο Σεντάι. Ένας από τους πιο φιλόδοξους στόχους μας ε, είναι ακριβώς αυτά να τα πετύχουμε και στην Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη. Συνάδελφοι, τελευταία μου παρατήρηση για την Παγκόσμια Ανθρωπιστική Σύνοδο. Αυτή η σύνοδος είναι πραγματικά μια ευκαιρία που παρουσιάζεται μια φορά σε μια ολόκληρη γενιά. Εν δυνάμει μπορεί να αλλάξει τελείως το τοπίο και την εικόνα της, ε, του όλου τοπίου για, την, για το σύστημα παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας. Θέλω και πάλι να ευχαριστήσω την Επιτροπή τη δική σας, την Επιτροπή Ανάπτυξης για τη βολή τη προ την Παγκόσμια Σύνοδο. Ιδίω ε, τον συνάδελφο σα Ερήγε Γκερέρο Σαλόμ για την έκθεσή του και γιατί όλα αυτά συνεισέφεραν στο να καθορίσουμε τη δική μας θέση και τοποθέτηση στην Παγκόσμια Σύνοδο, την Ευρωπαϊκή θέση. Ένα δεύτερο, μια δεύτερη φάση των συμπερασμάτων του Συμβουλίου θα εγκριθούν τον Μάιο. Αυτά θα επιβεβαιώσουν τις κοινέ μας δεσμεύσεις να κάνουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε για να πετύχουμε αποφασιστική δράση και μεταμόρφωση του ανθρωπιστικού συστήματος. Ε, εν ώψη της ε, Συνόδου το θεματολόγιο για την ανθρωπότητα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ θέτει ένα σαφές πλαίσιο για την ανάληψη δράσης. Πρόθεσή μου είναι να λάβουμε σοβαρότατες δεσμεύσεις στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ μαζί με τους συναδέλφους μου Μίμητσα και Γεωργίευα θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είναι ευθύνη όλων μας και είμαστε και από τους μεγαλύτερους δωρητές. Πρέπει να πιέσουμε τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Προσωπική μου άποψη, όπως ξέρετε, ήταν ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να περιχωρήσουμε σε μια πολιτική δήλωση, όμως τώρα συνειδητοποιώ ότι υπάρχουν δυσκολίες ως προς αυτή την επιλογή. Πολλές δυσκολίες. Πάντως, οι πολιτικές δεσμεύσεις είναι το ίστατο πλαίσιο προκειμένου να πετύχουμε συγκεκριμένα χειροπιαστά αποτελέσματα από, αυτό αυτή τη μεγάλη εκδήλωση, το μεγάλο γεγονός. Οπωσδήποτε θέλουμε ένα αποτελεσματικότερο σύστημα ανθρωπιστική βοήθεια. Οι ανθρωπιστικοί φορεί πρέπει να αναλάβουν δεσμεύσει, να συνεργάζονται καλύτερα, με κοινέ αξιολογήσει και σύστημα παρακολούθησης και με, λιγότερες, ε, με λιγότερο γραφειοκρατικό άκτο. Οι δωρητέ πρέπει να αναλάβουν και αυτοί το δικό του ρόλο και τι δικέ του ευθύνε. Θα μπορούσε αυτό να πάρει τη μορφή ενός, μια μιας μεγάλης ε, συμφωνίας. Νομίζω η Κωνσταντινούπολη είναι το καλύτερο μέρο για να πετύχουμε την επίτευξη αυτή τη συμφωνία. Πρέπει όμως να εργαστούμε σκληρά για να προλάβουμε και να επιλύσουμε τις διαφορές και ε, κατά κύριο λόγο να προωθήσουμε το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Με τεράστια άσκηση πιέσεων σε όλες τις κρίσεις. Ξέρετε, το πρόβλημα πλήττει τις ιατρικές ε, υποδομές και το προσωπικό σε πολλές χώρες και πολύ άσχημα. Θα ήθελα να επαναλάβω για την επιτυχία αυτής της Συνόδου χρειαζόμαστε αυθεντικές πολιτικές δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Είναι πραγματικά αρκετά σημαντικό. Είναι προϋπόθεση για να επιτύχουμε. Η Σύνοδος θα λήξει επισήμως στις 24 Μαΐου. Αλλά δεν θα είναι αυτό το τέλος της προσπάθειας. Θα είναι η αρχή. Η αρχή μιας εντατικής δουλειάς για να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις που θα αναλάβουμε στην Κωνσταντινούπολη. Το να δώσουμε συνέχεια στα αποτελέσματα της Συνόδου θα είναι κέρια προτεραιότητα για μένα και πιστεύω για όλους μας. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την υλοποίηση της ευρωπαϊκής ε, κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια το αποτέλεσμα της παγκόσμιας ανθρωπιστικής συνόδου, οι δεσμεύσεις που θα αναλάβουμε, όλα αυτά θα απεικονιστούν στο έργο μας. Φίλοι μου, και πάλι σας ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση. Αν υπομονώ να ακούσω τις απόψεις σας και τις προτάσεις σας, αλλά και τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Όταν ε, γίνατε Επίτροπος, αρχίσαμε με μια σειρά καταστροφών. Η κυρία Γιώργη έτσι έλεγε και τώρα τα πράγματα χειροτερεύουν. Η Εμένη για παράδειγμα είναι κάτι τρομερό. Κρίσεις που διαβάζουμε στις εφημερίδες Συρία, οι συγκρούσεις επαναλαμβάνονται και προστίθεται η μία στην άλλη. Μαρίκε Γκερέρο, Νταβοστήρ, Μαρί Χάουαρκ, ο κύριος Κούλογλου επίσης. Ποιος άλλος? Ο κύριος Βένσα. Για να ξέρουμε. Λοιπόν, έχουμε 35 λεπτά. Νομίζω ότι φτάνει ο χρόνος. Τρία λεπτά ο καθένας περίπου, έτσι. Ερίκη Γκερέρο πρώτα. Ναι, θα είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος, λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλά από αυτά που εγώ θα έθετα στον Επίτροπο, μας τα είπε ήδη ο από μόνος του. Τον ευχαριστώ λοιπόν, τον ευχαριστώ για το έργο του, για τη δουλειά που κάνει δηλαδή η Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ. Τον ευχαριστώ για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται σε έκτακτες περιστάσεις, τόσο μέσα όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον ευχαριστώ για αυτά που κάνει για τους πρόσφυγες, για παράδειγμα, για το παιδί. Και τον ε, ευχαριστώ και για τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις ε, φυσικές καταστροφές, τις θεομηνίες. Εκουαδόρ, για παράδειγμα, η σημερινός που περιμένει βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από τον τελευταίο σεισμό. Τον ευχαριστώ επίσης και για την δέσμευση που έχει αναλάβει όσον αφορά την εκπαίδευση. Αυτό αποτελεί μια ποιοτική αλλαγή στην έκτακτη βοήθεια. Επί τέσσερα έχει πολλαπλασιαστεί ο προπολογισμό για την εκπαίδευση. Το αναγνωρίσατε κι εσείς ότι σε αυτό βοήθησε πολύ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Για του χρόνου τώρα. Όσον αφορά το διαρθρωτικό διάλογο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του χρόνου είναι μια χρονιά που θα εκτιμήσουμε τι έχουμε κάνει με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει μέχρι τώρα στις διεθνείς διασκέψεις κατά τη διάρκεια του 2015. Θα αξιολογήσουμε δηλαδή τα αποτελέσματά μας στην Κωνσταντινούπολη. Πρέπει επίσης να αποφεληθούμε μαζί από κοινού. Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Επιτροπή Ανάπτυξης Κοινοβουλευτική να δούμε τι θα γίνει με τις δημοσιονομικές προοπτικές γιατί η συζήτηση από αυτών θα αρχίσει σύντομα. Θα δούμε λοιπόν πώς θα αναθεωρηθούν, γιατί από αυτό θα εξαρτηθούν και οι επόμενες δεσμεύσεις που θα αναλάβουμε, αλλά και οι πληρωμές που θα κάνουμε στην ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτά τα οποία θέσατε ως προτεραιότητα, η εκπαίδευση, ο εκτοπισμός, η αντοχή, ο ανθρωπιστικός νόμος, Όλα αυτά είναι πράγματα που ενδιαφέρουν πάρα πολύ την Επιτροπή μας, ιδιαίτερα το τελευταίο για το International Humanitarian Law. Πολλές επιθέσεις γίνονται τελευταία. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνει συζήτηση μετά από πρωτοβουλία της δικιάς μας Επιτροπής την επόμενη εβδομάδα επί τη ευκαιρία ενός ψηφίσματος που θα εγκρίνουμε. Στην ομάδα μου γνωρίζετε, και το γνωρίζετε γιατί σας το έχουμε πει, ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε τη συνέχεια του προγράμματος δράσης για την Ευρωπαϊκή Συνένεση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Εκπνέει του χρόνου, το 2017. Θέλουμε λοιπόν να δοθεί συνέχεια. Επίσης, η ομάδα μας ενδιαφέρεται πολύ για να εξετάσει τις ιδιαιτερότητες της κάθε κρίσης μεγάλης διάρκειας και θέλουμε να ενισχύσουμε τις τοπικές δυνάμεις προκειμένου να βοηθήσουν να ξεπερνιόνται οι κρίσεις. Κάτι τώρα για την ανθρωπιστική διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης. Πρώτον, τι είναι το σημαντικό. Καταλαβαίνω ότι πράγματι το σημαντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να πάει εκεί με συγκεκριμένες δεσμεύσεις εύστοχες πολιτικά με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Τόσο λοιπόν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαΐου, όπως και οι δεσμεύσεις που ανακοινώθηκε ότι θα αναλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το σημαντικό επί τη ευκαιρία της διάσκεψης αυτής. Και το δεύτερο είναι ότι στις 24 του μηνός δεν τελειώνουν τα πράγματα. Από τους 24 του μηνός και μετά πρέπει να φροντίσουμε ότι οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει θα υλοποιηθούν. Υπάρχει και ένα μικρότερο πρόβλημα, αλλά είμαι υποχρεωμένος να το θέσω. Ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας που θα πάει στην Κωνσταντινούπολη, έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα παρουσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις συζητήσεις της Κωνσταντινούπολης και της Κομισιόν φαντάζομαι επίσης. Γιατί δημιουργήσαμε μία αντιπροσωπεία με 11 μέλη και τελικά δεν γνωρίζουμε ούτε καν αν τέσσερις θα πάνε ή δύο θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο σύνολο των συζητήσεων. Οι υπόλοιποι θα συμμετάσχουν σε διασκέψεις, σημαντικές ομάδες εργασίας, αλλά όχι παντού. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, απλώς να τονίσω ότι θεωρώ ότι είμαι υπεύθυνο και για τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν όσο γίνεται περισσότερο. Γι' αυτό και ζητάω ό,τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας βοηθήσει να το κάνει. Και ώστε οι προσκλήσεις να είναι πιο ουσιαστικές για συμμετοχή μας στις εργασίες στην Κωνσταντινούπολη και αυτό όχι μόνο για την ίδια την αντιπροσωπεία αλλά και για το επίπεδο του έργου μας όσον αφορά την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριο Στίερ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τον Επίτροπο. Τον ευχαριστώ για την ενημέρωσή του όσον αφορά τις διάφορες κρίσεις που αντιμετωπίζουμε. Και πάνω απ' όλα τον ευχαριστώ πολύ για το έργο του. Ξέρετε Επίτροπε, ότι μπορείτε να βασιστείτε στη στήριξη της δικιάς μας ε, πολιτικής ομάδας και θα συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε. Έχουμε δει πραγματικά βελτίωση σε πολλούς τομείς. Ο Ενρίκε ήδη το είπε και εσείς έχετε αναφερθεί στην εκπαίδευση. Όντως, εκεί υπάρχει βελτίωση. έχετε πει ότι είναι από τις πρώτες προτεραιότητές σας. Τώρα γενικότερα για τις προτεραιότητες στο διευθυντικό διάλογο, το μήνυμά μας είναι η σημασία που έχει η συνέχεια και η ενίσχυση θα έλεγα της ανακούφισης με την ανάπτυξη. Ανθρωπιστική βοήθεια δηλαδή, αλλά και αναπτυξιακή αρρωγή η σχέση αυτών των δύο θα έπρεπε να ενισχυθεί περισσότερο. Και θα ήθελα να ξέρω περισσότερα για δράσεις ή σχέδια που έχετε υπόψη σας επ' αυτού. Ένα συγκεκριμένο τομέα, βέβαια, είναι η εκπαίδευση, όπως είπαμε. Επιπλέον από την αύξηση του προπολογισμού, ένα άλλο ζήτημα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι και ανάπτυξη συγκεκριμένων πολιτικών για την εκπαίδευση. Αυτό θα το συζητήσουμε με τους συναδέρφους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για το μελλοντικό έργο της Κομισιόν. Όταν μιλάμε για πολιτικές, η εκπαίδευση είναι κάτι που μπορούμε να δούμε με διαφορετικές διαστάσεις στα πλαίσια της ανθρωπιστικής κρίσης. Πρέπει να δούμε ποιοι είναι εταίροι μας επιτόπου οι διεθνείς οργανώσεις που μερικές φορές μπορούν να έχουν περισσότερο πρόσβαση. Μερικές φορές πάλι είναι ένα ευαίσθητο θέμα γιατί ακριβώς οι ίδιες αυτές οι οργανώσεις μας έχουν πει ότι θα θέλαν να καταλάβουν καλύτερα ακόμα πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλο πάντων, θα πρέπει να αναλύσουμε περισσότερο αυτές τις πολιτικές και ίσως να σκεφτούμε νέες κατευθυντήριες γραμμές. Επιπλέον, πώς αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις της νομοθεσίας για την ανθρωπιστική βοήθεια. Ξέρω ότι και άλλοι συνάδελφοι θα αναφερθούν σε αυτό. Απλώς τονίζω ότι και για τη δικιά μας την ομάδα το ΕΛΚ είναι ένα σημαντικό θέμα. Τέλος, αναφερθήκατε στη δύσκολη κατάσταση στην Ιεμένη. Είπατε ότι πήγατε και στο Ιράν. Στην Ιεμένη, όπως και στη Συρία, υπάρχει πόλεμος διανταποκρίσεως. Πώς εκτιμάτε τη συνεργασία της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράν, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση της βοήθειας. Είναι κάτι που συζητήσατε κατά την επίσκεψή σας εκεί. Ευχαριστώ. Η Μαρία Χόιπουκ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ε, Επίτροπε που έρχεστε τακτικά πάντοτε και έχετε τακτικές ανταλλαγές απόψεων μαζί μας. Μιλήσαμε ήδη για αυτή την χρηματοδότηση και την καλύτερη σύνδεση της άμεσης βοήθειας με την πιο μακροπρόθεσμη βοήθεια. Και εγώ βλέπω κάποιο δυναμικό εδώ να υπάρχει. Υπήρχαν κάποια ελλείμματα ή κάποια αναντιστοιχεία μεταξύ των αναγκών ανθρωπιστικής βοήθειας επειδή είναι πολλές οι κρίσεις πια σήμερα, και των κονδυλίων που όντως διατίθενται. Γιατί η αύξησή τους προβλέπεται σε πολύ περιορισμένα μονοπλαίσια. Και Πιστεύω ότι η συνεργασία και η σύνδεση αναπτυξιακής με ανθρωπιστική βοήθεια θα πρέπει να γίνει ακόμη περισσότερο. Και εσείς ο ίδιος μας δώσατε σχετικά παραδείγματα και θα με ενδιέφερε να μου πείτε αν βλέπετε κάποια πρόοδο εδώ ήδη να έχει σημειωθεί ή είμαστε ακόμα στην αρχή. Επίσης ε, υπάρχουν σχέδια στα πλαίσια της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας που αντικατοπτρίζονται και συμπεριλαμβάνονται στο πολιετές δημοσιονομικό ε, πρόγραμμα και μπορούν έτσι να εξεταστούν. Κάτι άλλο που μας είπατε είναι ότι στα πλαίσια της ανθρωπιστικής βοήθειας οι οργανισμοί επιτόπου πρέπει, οι οργανώσεις, πρέπει να συνεργάζονται καλύτερα. Ε, και θα με ενδιέφερε να δω πώς το βλέπετε εσείς, πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις. Γιατί και εδώ χρειάζεται μια ανάλογη οργάνωση. Και μια και μιλάμε για τη χρηματοδότηση, ένα τελευταίο. Η σύνδεση της ανθρωπιστικής με το, την COP21. Εσείς μιλήσατε για τις επώδυνες ε, εμπειρίες που είχατε στην Αιθιοπία ο Ελνίνιο είναι κομμάτι της κλιματικής αλλαγής και επειδή μιλήσατε για πρόσθετα κονδύλια, αυτά από πού θα βρεθούν, πρέπει δηλαδή να βρεθούν κάπου αλλού από την αναπτυξιακή βοήθεια ή θα δημιουργηθούν κονδύλια για κλιματικά προβλήματα που στο μέλλον θα είναι περισσότερα. Δηλαδή μιλάμε για συμπληρωματικό προϋπολογισμό, πρόσθετα χρήματα. Ε, αυτό ίσως θα ήταν αναγκαίο. Και το τελευταίο θέμα, η παραβίαση του ανθρωπιστικού δικαίου, όλο και περισσότεροι ε, εμπλεκόμενοι ε, κινούνται σε σημεία κρίσεων, ε, είναι επικεφαλής αντιπαραθέσεων και σημειώνονται πολλές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Σκεφτείτε το βομβαρδισμό των εγκαταστάσεων των γιατρών χωρίς σύνορα. Υπάρχουν πρωτοβουλίες που μπορείτε εσείς να αναλάβετε για να αντιμετωπίσετε αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα. Γιατί τι να τα κάνουμε τα λεφτά αν δεν υπάρχει πρόσβαση εξασφαλισμένη για τις οργανώσεις μας, για τις εγκαταστάσεις μας, ούτω ώστε να βοηθήσουν επί τόπου. Άλλη μια φορά ένα θερμό ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Ευχαριστώ Μαρία. Ο κύριος Κουλόγλου. Ε, ε, ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την ενημέρωση. Ήθελα να σας ε, υποβάλω δύο ερωτήματα και να κάνω και μια πρόταση. Το πρώτο ερώτημα είναι ε, ότι Πράγματι έγινε σε χρόνο ρεκόρ η εκταμίευση των πρώτων ποσών. Αυτά τα ποσά πήγανε στην ε, ανώτατη ε, αρμοστία του ΟΗΕ για τους ε, πρόσφυγες, τον, ε, επίσης τον Ερυθρό Σταυρό και σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Στο ίδιο διάστημα όμως, το ελληνικό κράτος ξοδεύει χρήματα. Ο στρατός δίνει το φαγητό, ε, οι τοπικοί δήμαρχοι δίνουν επίσης εγκαταστάσεις και εξοδεύουν χρήματα για να φτιάξουν στρατόπεδα. Τα νοσοκομεία δίνουν ε, επίσης ε, χρήματα και ξέρετε ότι λόγω της κρίσης και της λιτότητας πολλά νοσοκομεία στην Ελλάδα είναι ήδη στα όρια. Δεν έχουν ούτε θερμόμετρα. Άρα ε, αναρωτιέμαι εάν ε, σχεδιάζεται ένα μέρος των ποσών αυτών ε, να δοθούν στο ελληνικό δημόσιο ή στις τοπικές ε, αρχές και πόσο θα είναι αυτό το ποσό. Το, η δεύτερη ερώτηση που είχα να σας κάνω. Προχτές την Κυριακή πήγα σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στον Κατσικά, είναι ε, στο, στα Ιωάννινα, ε, σε μια πόλη που είναι στα βορειοδυτικά της Ελλάδας. Η κατάσταση είναι δύσκολη, γίνονται βελτιώσεις, αλλά είναι δύσκολη. Είδα ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά παιδιά. Και το ερώτημα είναι ε, αν θα μείνουν αυτοί οι άνθρωποι που μάλλον θα μείνουν για καιρό εκεί ε, τι θα γίνει με την εκπαίδευση των παιδιών ε, από τώρα και επίσης ε, από, τον, ε, από τον, τον ερχόμενο, την ερχόμενη σχολική χρονιά, από το Σεπτέμβριο. Είπατε ότι θα δώσετε κάποια χρήματα, γι' αυτό δεν κατάλαβα ακριβώς τα 44 εκατομμύρια που αναφέρατε, αλλά και θα είναι παραπάνω από τα 44 εκατομμύρια, ε, πόσα λεφτά θα είναι για την εκπαίδευση και πότε θεωρεί ότι θα, θα, εκταμιευθούν. Είναι. Και τελειώνω με την πρόταση που είχα να σας κάνω. Κοντά στο στρατόπεδο αυτό υπάρχει ένα παλιό ορφανατροφείο, πολύ μεγάλο, το οποίο πλέον δεν λειτουργεί. Αλλά είναι σε καλή κατάσταση είναι σε εξαιρετικό μέρος, ιδηλιακό μέρος ε, και έχει όλες τις εγκαταστάσεις. Και θα σας πρότεινα, δίνοντας στον κατάλληλο φορέα τα χρήματα που αναλογούν, να κάνετε αυτό το κέντρο πρότυπο προσφυγικό κέντρο, να το βάλετε υπό την εποπτεία της δικής σας ή της Επιτροπής μας, της ΔΕΒΕ ή και το δύο μαζί και να το κάνουμε πρότυπο κέντρο για να δείξουμε μια άλλη εικόνα σε όλο τον κόσμο για το πώς η Ευρώπη μπορεί να μεταχειριστεί τους ανθρώπους αυτούς που είναι σε ανάγκη. Ευχαριστώ. Um, thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Πέντερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Από αυτά που μας είπατε, δείξατε ότι σβήνεται μια φωτιά και αμέσως πιάνει μια νέα πυρκαγιά. Αναφερθήκαμε στην εκπαίδευση. Πολλοί συνάδελφοι το είπαν όντως. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό για όλους μας. Το ξέρουμε ότι στους καταβλισμούς υπάρχουν οικογένειες με παιδιά που συχνά χρόνια περνάνε σε τέτοιους καταβλισμούς, μεγαλώνουν τα παιδιά στους καταβλισμούς. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, χρειάζονται εκπαίδευση. Αν δεν τους δώσουμε τα μέσα, τότε ριζοσπαστικοποιούνται. Άρα, διακινδυνεύει η ασφαλειά μας. Ρωτάω λοιπόν, έχετε τίποτα προγράμματα, υποτροφίες για παράδειγμα για τους νέους αυτούς που να μπορούν να βγουν από τους καταβλισμούς, να παίρνουν υποτροφίες και να μπορούν να είναι υποψήφιοι. Μερικές φορές όταν απορριφθεί μια φορά η αίτησή τους δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν νέα. Αυτό οδηγεί σε απογοήτευση. Οπότε αυτά που μας είπατε εδώ ότι θέλετε να στηρίξετε την εκπαίδευση θέλω να ξέρω με ποιο τρόπο. Πρέπει να έχουν κίνητρα. Οι νέοι αυτοί που ζουν στους καταβλισμούς φτάνουν παιδιά και μεγαλώνουν εκεί. Ευχαριστούμε. Τελευταία ερώτηση. Μπέτρις Μπεσέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που πάντα είσαστε στην διάθεσή μας και όντως εσείς μας δίνετε αυτή την εικόνα των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά θέλω να αναφερθώ σε αυτά και στις πληροφορίες που μας δίνετε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και γιατί βρίσκω γενικά ενδιαφέρον το θέμα, αλλά και γιατί εγώ ασχολούμαι όλους ιδιαίτερος με αυτά. Δεν θα επαναλάβω αυτά που ρώτησαν οι συνάδελφοι. Εγώ όμως θέλω να πω ότι η άμεση αντίδραση είναι πολύ σημαντική αρχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προσθέτη αξία. Είτε πρόκειται για τα παιδιά, είτε πρόκειται για τα κονδύλια για την Ελλάδα. Είδαμε πως εσείς προσωπικά συμμετάσχατε. Όσον αφορά τώρα τις ανθρωπιστικές κρίσεις, είναι κοντά μας, όλο και πιο κοντά μας και είναι όλο και πιο μεγάλες. Είδαμε ότι πήγατε και στην θα ήθελα να ξέρω μάλλον για τη Βενεζουέλα. Δεν έχει καθόλου φάρμακα. Εκτός από την έλλειψη τροφίμων, πρόσβαση σε νερό. Φαίνεται ότι η κατάσταση θα είναι κρίσιμη εκεί και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε. Γιατί και η πολιτική κατάσταση είναι δύσκολη εκεί. Θέλω να σας μεταφέρω το ενδιαφέρον που πρέπει να δείξουμε στην εκπόνηση αυτής της νέας Ευρωπαϊκής Συνένεσης για την Ανάπτυξη. Μιλήσαμε γι' αυτό σήμερα το πρωί στην Επιτροπή μας. Είμαστε σε μια σημαντική στιγμή. Έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας πολλά πράγματα. Η ανθρωπιστική βοήθεια και η αναπτυξιακή βοήθεια πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι οι κρίσεις που κρατούν πολύ καιρό, είτε πρόκειται για τη Σαχάρη, είτε για το Λίβανο, είτε οπουδήποτε αλλού, απαιτούν να έχουμε πάντα υπόψη μας και την ανάπτυξη συγχρόνως. Και η ανθρωπιστική βοήθεια με την ανάπτυξη πρέπει να αποτελούν τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, για να οικοδομήσουμε μια κοινωνία περισσότερο ισότιμη, με πολίτες που είναι ίσοι μεταξύ τους. πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και μία βιώσιμη έννοια για την ασφάλεια. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στην γενική μας στρατηγική. Όπως έχουμε ήδη πει, τα σχολεία, τα νοσοκομεία χρειάζονται στήριξη. Όσοι δουλεύουν στις διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις χρειάζονται τη στήριξή μας. Για να έχουμε ασφάλεια πρέπει να έχουμε και την ευκαιρία να είναι βιώσιμοι οι στόχοι του 2030. Άρα, ισότητα, εκπαίδευση, χρηστή διακυβέρνηση, αλλά και υγεία. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Και τέλος, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι και η μετανάστευση μπορεί να είναι και κάτι θετικό, δεν είναι μόνο κρίση. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σήμερα το πρωί οι συντονιστές μιλήσαμε για το κατά πόσο θα υπάρχει νέα συνένεση για την ανθρωπιστική βοήθεια μετά τη διάσκεψη. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη από αυτού, αν πιστεύετε ότι θα ήταν χρήσιμο. Σε εσά ο λόγος τώρα. Επιτρέψτε να ξεκινήσω το θέμα που ήγερε ο, ο καλός μου συνάδελφος και φίλος Ενδύε Κεραίρο Σαλό σχετικά με το World Humanitarian Summit και τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, όχι μόνο επικροτώ τα όσα είπες, αλλά πιστεύω ακράδαντο ότι η δική σας παρουσία εκεί δεν θα είναι απλώς ενισχυτική για την ευρωπαϊκή παρουσία, αλλά θα είναι και βοηθητική για τα ίδια τα αποτελέσματα της Συνόδου, γιατί προσκομίζεται κάτι διαφορετικό που έχει σχέση με την ίδια την κοινωνία των πολιτών και θα έρθετε σε επαφή με τη μεγάλη συμμετοχή εκεί σε αυτό το μεγάλο event. Ε, Ασχολήθηκα με το θέμα εδώ και δύο μήνες. Βλέπω πρακτικές δυσκολίες από, τον, από πλευράς Ηνωμένων Εθνών και από πλευράς φιλοξενούσας χώρας που είναι η Τουρκία. Βέβαια όλα αυτά ανάγονται στο επίπεδο του προβλήματος της ασφάλειας, του security. Οι τελευταίες μου επαφές και με τους Τούρκους συναδέλφους είναι ότι επειδή δεν μπορούν μέχρι τώρα να αξιολογήσουν τη συμμετοχή σε ανώτατο επίπεδο ηγετών. Γι' αυτό ε, ακόμα και στα ξενοδοχεία έχουν κατά κάποιο τρόπο ζητήσει να κλειστούν υπηρεσίε ζωμάτια που μπορεί στο τέλο να μην χρειαστούν, γιατί δεν θα υπάρχει αυτή η συμμετοχή. Και εκεί μπορούν να κάνουν αναπροσαρμογή τη μέχρι τώρα τακτική και στρατηγική. Ελπίζω μέσα σε αυτή την αναπροσαρμογή να μπορέσω και εγώ προσωπικά να βοηθήσω έτσι ώστε η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετάσχει ακόμα περισσότερο στις εργασίες της Συνόδου στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Θα κουβεντιάσω το θέμα αύριο το πρωί φεύγω για τη Νέα Υόρκη για συναντήσεις για το WHS και θα έχω συνάντηση με τον Στίβεν Ομπράια και θα το, το συζητήσω μαζί του ειδικά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το πιστεύω ότι χρειάζεται να αναβαθμιστεί η παρουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, όπως πάντα. Και ακριβώς επειδή και στις προσωπικές μας συναντήσεις βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους και συζητάμε πάρα πολύ ανοιχτά και καθαρά και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε αυτόν τον ειλικρινή διάλογο. Και έχεις απόλυτο δίκαιο ότι με το WHS και στις 24 του μήνα αρχίζει πιο μεγάλο έργο διότι θα είμαστε αναγκασμένοι αυτά που θα συμφωνήσουμε να εφαρμόσουμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απολύτως ότι θα πρέπει στο διαρθωτικό διάλογο και στην αξιολόγηση των δημοσιονομικών προεπτικών να βρούμε λύσεις μέσα από τις πρώτες αξιολογής που θα κάνουμε. Σε ό,τι αφορά το consensus, σχεδιάζουμε μια έκθεση προόδου για το implementation plan during the, κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας, στο επόμενο εξάμεινο, και είναι πολύ σημαντικό. Κάτι που αφορά το Σεντάι και την εφαρμογή του Υπάρχει ένα σχέδιο δράσης που θα δημοσιοποιηθεί, δημοσιο, δημοσιοποιηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Να πω κάτι για τον κανονισμό και όπως είπα και πριν στην εισαγωγή μου θα το δούμε σε σχέση με τα αποτελέσματα του WHS. Και μια και αναφερθήκαμε τόσο στο θέμα του Education Emergencies να πούμε ότι θα έχουμε μια αξιολόγηση η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και ελπίζω να είναι έτοιμη το τρίτο εξάμεινο, το τρίτο ε, τρίμηνο του, 2000, του παρόντος χρόνου. έχετε αναφερθεί πολύ στο θέμα της σύνδεσης του humanitarian phase με τον development phase. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι είναι μεγάλη πρόκληση. Εάν ισχυριστώ ότι με βάση την εμπειρία μου είμαι απολύτως ικανοποιημένος, θα είναι λάθος. Θεωρώ ότι έχουν πάρα πολλά να γίνουν σε αυτό τον τομέα. Και αν γίνουν πολλά, σε αυτόν τον νομέα θα μπορούμε ενδεχομένως να περιορίσουμε και κόστος και να, μεταφέρουμε λεφτά σε άλλες περιοχές για να γίνουμε πιο efficient και πιο effective. Όμως, έχουμε ήδη κάποια θετικά αποτυπώματα στην εφαρμογή, παραδείγματος χάρη, του Education in Emergencies στην Τουρκία όπου τα προγράμματα για το informal education συνδέονται με τα προγράμματα που προσφέρει η Indigenia, έχουν αποκτήσει αυτό το χαρακτήρα της σύνδεσης. Τα δικά μας προγράμματα από το Humanitarian Assistance που εξειδικεύονται στο informal education δημιουργούν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτοί οι μαθητές να μπορούν να μπουν στο formal education. Και όπως το ήρε και ο κύριος Βέτα, είναι, προετοιμάζουμε για να είναι μέσα στα πλαίσια ενός curriculum που θα τους οδηγεί ακόμα ενδεχομένως και στις εξετάσεις για πανεπιστήμια. Και εκεί βέβαια θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο υποτροφιών, όπως πολύ ίσως τα είπατε, για να δίνουμε ελπίδα και προοπτική γιατί τα παιδιά θέλουν ελπίδα και προοπτική. Και συμφωνώ απολύτω με τη θέση που καταγράφηκε την, και το είδα on the ground στην Κένια, στο Τατάπ camp ότι εάν δεν υπάρχει ελπίδα και προοπτική, και αν δεν υπάρχει συνέχεια στην εκπαίδευση είναι η βάση για το radicalization. Είναι γι' αυτό που έδωσα μεγάλη έμφαση και ε, έκανα ως προτεραιότητά μου το education emergency. Ήταν η εμπειρία που βγήκε on the ground. Δεν ήταν μια θεωρητική σκέψη η οποία εμφανίστηκε έτσι out of the blue. Θέλω να απαντήσω ειδικά στον συνάδελφο κύριο Κούλογλου για τα θέματα που έθεσε, διότι κάποια από αυτά τα κουβέντιασα και χθε στην Αθήνα με τον Υπουργό Μετανάστευση, τον κύριο Μουζάλα, ένα πολύ αξιοπρεπή άνθρωπο και φωσιωμένο στη δουλειά που κάνει. Και τα κουβέντιασα και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρο. Οι διευκρινήσει είναι οι εξή. Τα λεφτά της ανθρωπιστικής βοήθειας ποτέ δεν διοχετεύονται μέσω κρατικών καναλιών. Αυτό είναι αρχή. Πάντα διοχετεύονται μέσω των humanitarian partners on the ground. Που σημαίνει αυτά τα λεφτά που ήδη αποφασίσαμε για την έκτακτη βοήθεια και αυτή τη στιγμή η χώρα η οποία εκπληρεί προϋποθέσεις για να παίρνει αυτή τη βοήθεια είναι η Ελλάδα, θα πάνε μέσω ανθρωπιστικών οργανώσεων. Και αυτά τα πρώτα 83 εκατομμύρια που υπογράψαμε τρεις μέρες μετά την απόφαση του Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, τέσσερις μέρες, πόσες ήταν, είναι μέσω ανθρωπιστικών οργανώσεων. Όλα. Όμως, ξέρουν όλοι πολύ καλά ότι υπάρχουν κι άλλα πολλά ευρωπαϊκά ταμεία από τα οποία μπορούν να πάρει λεφτά η ελληνική κυβέρνηση να αξιοποιήσει έτσι ώστε να δημιουργήσει υποδομές και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Είτε μέσω του Migration Fund, είτε IHS που είναι υπεύθυνο ο Δημήτρης Αβραμόπουλο. Αύριο θα είναι στην Αθήνα η Επίτροπος Μάριαν Τάισεν ακριβώς για να συζητήσει αξιοποίηση από κονδύλια social affairs. Που σημαίνει υπάρχει μια ευρία γκάμα δυνατότητας αξιοποίησης ευρωπαϊκών ταμείων που αφορούν και τους Έλληνες πολίτες και τους πρόσφυγες σε αυτή την κατεύθυνση. Τα λεφτά της ανθρωπιστικής βοήθειας πάνε μέσω των ανθρωπιστικών οργανώσεων. Έχουμε όμως συμφωνήσει για όλα τα project να είναι, και εδώ είναι η διαφορά ενός member state από χώρες της Αφρικής ότι θα είναι in coordination, in cooperation with the member state, με την Ελλάδα, με τα Greek authorities, με την ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό συμφωνήθηκε στη συνάντηση που είχαμε με τους humanitarian partners και τον Υπουργό Μετανάστευση. Που σημαίνει είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η συνεργασία να αποτυπωθεί στην πράξη και το κλίμα που είδα χθε στην Αθήνα ήταν εξαιρετικό. Και γι' αυτό ευχαρίστησα τον κύριο Μουζάλα που θα βοηθήσει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Διευκρίνηση γιατί θα είναι πέραν των 52 εκατομμυρίων που αφορά και άλλους. Τα 52 εκατομμύρια είναι το αποτέλεσμα της αύξησης του στόχου από το 1% στο 4%. Στην Ελλάδα όμως υπάρχουν κονδύλια για education in emergencies μέσα σε αυτά τα 83 εκατομμύρια που είναι από άλλη πηγή, που σημαίνει είναι πέραν των 52 εκατομμυρίων. Και για την Τουρκία, αυτή τη στιγμή, επειδή υπάρχει το Turkey Facility, τα λεφτά για το education είναι πέραν των 52 εκατομμυρίων που προέρχονται από το 1 δισεκατομμύριο που έχουμε για ανθρωπιστική βοήθεια από τα 3 δισεκατομμύρια μέσα στην Τουρκία. Κάποια από αυτά τα λεφτά, ήδη 45 εκατομμύρια, έχουν υπογραφή συμβάσει για το education emergency, informal education και είναι πέραν των 52 εκατομμυρίων. Που σημαίνει ότι τελικά εάν αθροίσουμε το συνολικό ποσό για το education για αυτό το χρόνο θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 50-52 εκατομμύρια που ήταν ο δικός μας στόχος διότι παίρνουμε από διαφορετικές πηγές. Σε ό,τι αφορά την πρότασή σας για τον Κάτσικα και το ορφανοτροφείο. Ε, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια προσπάθεια και με άλλους επιτρόπους, μέσα από άλλα φαντς τα οποία μπορούν να κάνουν την αποκατάσταση αυτού του χτιρίου που λέτε του ορφανοτροφείου, να το κουβεντιάσουμε μετά και με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο που έχει αυτά τα λεφτά και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό ακριβώς να γίνει πρότυπο και μια επίσκεψη από κοινού θα ήταν καλή στην περιοχή και στο συγκεκριμένο καταβλισμό για να του δείξουμε ακριβώς την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και το ότι υπάρχει μια ποιοτική διαχείριση του προσφυγικού. Γιατί αυτό είναι ένα στίχημα και θα πρέπει αυτό το στίχημα να το κερδίσουμε. Uh, Θα σας δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο, μην ανησυχείτε. Ευχαριστώ πολύ. για τις παραβιάσεις του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου. Για το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Ότι δεν είναι δυνατόν να ανεχτούμε ως ανθρωπιστική οικογένεια να δέχονται χτυπήματα νοσοκομεία, νοσοκόμοι, νοσοκόμες και humanitarian workers. Προσωπικά πίστευα και πιστεύω ότι πρέπει μέσα από το WHS να κερδίσουμε ένα political commitment ότι θα υπάρχουν κυρώσεις σε χώρες που χτυπούν humanitarian workers και νοσοκομεία και άλλα, άλλες εγκαταστάσεις ανθρωπιστικών οργανώσεων. Είναι ψηλό στόχος, αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον στην Κωνσταντινούπολη ας ξεκινήσει η συζήτηση. Και δημιουργεί, εν πάση περιπτώσει, ένα πολιτικό κλίμα που ο κάθε ένας θα μπορεί να σκέφτεται διπλά πριν κάνει την οποιαδήποτε επιχείρηση απέναντι σε στόχου που δεν ξέρει. Γιατί πολλέ φορέ μπορεί να γίνει από Αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία είχε να είσαι πάρα πολύ προετοιμασμένο. Ακόμα και σε περιόδου πολέμου. Ε, θέλω να εντοπίσω τη συζήτηση στο ρόλο των host communities και των local actors. Υπόθηκε και από εσά και είναι πάρα πολύ σωστή. Η εμπειρία μου είναι ότι εάν δεν υπάρχει ενεργοποίηση των local actors, τελικά και η ανθρωπιστική βοήθεια και η αναπτυξιακή βοήθεια έχουν ένα μεγάλο κενό. Και Χθες στην Ελλάδα, στη συζήτηση που κάναμε και ήταν μια συζήτηση που ακολούθησε την παρουσία του Φιλίππο Κράντι στο Foreign Affairs ε, ε, Council όπου το UNHCR δεσμεύτηκε ότι θα αξιοποιεί πάρα πολύ τους λοκαλάχτους. Γιατί έχουν την εμπειρία και κυρίως μπορούν να συμφιλιώσουν τους, την κοινότητα των προσφύγων με τα host communities. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά στην Ελλάδα και στην Τουρκία, που το ζω διότι έχω επισκεφθεί πολλές φορές, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει αυτή η στήριξη των, του public opinion, των κοινωνιών. Και αυτή η στήριξη θα βασιστεί και στην αξιοποίηση των local actors αλλά και στο ότι θα γίνει κατά κάποιο τρόπο αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων. Από μια προσωπική μου εμπειρία στο Καζιάντεπ, επειδή χρησιμοποιήθηκε πολύ σωστά το σύστημα του cash and voucher, στο Καζιάντεπ η πόλη, οι κάτοικοι της πόλης αντιμετωπίζουν τους πρόσφυγες του Σύριου με έναν τρόπο πολύ πιο ανοιχτό γιατί και αυτοί έχουν κάποιο κέρδο εξαιτία του cash voucher. Να είμαστε ρεαλιστέ στο πώ οι άνθρωποι πολλέ φορέ αντιμετωπίζουν αυτέ τι κρίσιμε καταστάσει. Και θυμάμαι ότι έμπαινα στα καταστήματα τα οποία ήταν συνδεδεμένα με το σύστημα cash and voucher και αντιμετώπιζαν τον Ευρωπαίο Επίτροπο, την Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου ως χορηγό. Διότι και αυτοί είχαν κάποιο κέρδο εξαιτία τη παρουσία. Θα μου πείτε αυτό ε, είναι μια πραγματικότητα η οποία βοηθά τουλάχιστον όχι μόνο να ανέχονται του πρόσφυγε, αλλά να νιώθουν ότι είναι μέρος της δική του κοινωνία. Είναι part of the integration τελικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη δούμε και σε αυτή τη διάσταση. να πω κάτι για το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία. Γιατί είναι, ήταν πολύ σημαντική επίσκεψη. Ε, οφείλω να πω ότι η, η πρωτοβουλία και η πολιτική εμπλοκή της ε, Φεντερίκας Μογκερίνη σε αυτό το θέμα του ντύλ με το Ιράν είναι αξιοσημείωτη και πιστεύω ότι βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρόλο της ως global actor. Το Ιράν μέσα από τις συζητήσεις που είχαμε δείχνει να θέλει να παίξει ένα θετικό ρόλο σε όλες τις κρίσεις στην περιοχή. Ακόμα και για την ΕΜΕΝ. Βοήθησε στο να υπάρχει humanitarian access για humanitarian βοήθεια στις αποκλεισμένες περιοχές της Συρίας μέσω κάποιων διασυνδέσεων που έχει και αυτό είναι σημαντικό και έδειξαν μεγάλη προθυμία στην αντιμετώπιση των Αφγανών προσφύγων. Εμείς αυξήσαμε τη βοήθεια, συζητήθηκα βέβαια και θέματα human rights, δεν υπάρχει αφιβολία. Δεν είναι κάτι που το κρύψαμε κάτω από το χαλί. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το κανάλι επικοινωνίας που άνοιξε θα είναι βοηθητικό και στην Ιεμένη η σύγκρουση μεταξύ Ιραν, Ιρανών και Σαουδάραμων στο θέμα είναι γνωστή, αλλά τουλάχιστον αυτή η επικοινωνία μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να το πρώτο βήμα που έγινε με την εγκεχηρία να δημιουργήσει την προϋπόθεση για το επόμενο βήμα και φαίνεται ότι οι Ιρανοί είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Μένουν πολλά να κρυθούν στην πράξη. Ευχαριστώ και πάλι. Θα πω τελικό τελική κουβέντα ότι όποτε έρθω στην Επιτροπή φεύγω σοφότερος. Γιατί αναγκάζομαι και εγώ να σκέφτομαι πράγματα τα οποία εγείρεται και να προσπαθώ να βρίσκω τις βέλτιστες δυνατές λύσεις. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Okay, well, thank, thank Επίτροπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Βέβαια, ε, όπως στη Γάζα βλέπουμε την ανάγκη και στην Ελλάδα σήμερα εκπαίδευση παιδιών, γιατί θα μείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από ό,τι φαίνεται. Αύριο στις 9.30, ακριβώς στις 9.30, θα είμαστε στην ώρα μας. Γιατί είναι και θέμα πρωτοκόλλου. Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε, που ήρθατε.